Mes chers collègues, bonjour à tous. Avant euh, d'entamer notre ordre du jour, euh, je voudrais euh, donc avoir. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε αυτό που έγινε τις τελευταίες ώρες στη Σομαλία, θανατηφόρες απόπειρες, τρομοκρατικές και οι οποίες θεωρούνται όπως είπα τρομοκρατικές ήδη. Η απειλή είναι γεωστρατηγικής εμβέλειας και πριν ξεκινήσουμε λοιπόν θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο τους νεκρούς αυτών των απαράδεκτων τρομοκρατικών ενεργειών και στη Σομαλία. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ και θα ξεκινήσουμε υποβάλλοντας προσέκριση την ημερήσια διάταξη την οποία λάβατε αν δεν υπάρχει διαφορετική άποψη θεωρείται δεκτή. Λοιπόν, η συνεδρίασή μας σήμερα θα είναι σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα μία ώρα και μισή ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση, τη λεπτομερή της πολιτικής ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης θα το αφιερώσουμε στην παρουσίαση της μελέτης για τις πολιτικές της Ένωσης στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συνοχή και αποτελεσματικότητα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο 2 είναι οι ανακοινώσει της πλευράς μου, δεν υπάρχουν ανακοινώσει. Θα συνεδριάσουν οι συντονιστές μετά τη συνεδρίαση και οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση. Τρίτο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής ασφάλειας. Θα γίνει μια παρουσίαση από πλευρά των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας το οποίο έχουμε, θα ξεκινήσουμε τον κύκλο ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την αξιολόγηση των νομοθετικών ρυθμίσεων, την παρουσίαση των ειδικών μέτρων, τα οποία λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αυτή η λεπτομερής αν θέλετε εξέταση θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε το τι υπάρχει σήμερα και στη συνέχεια να δούμε ποια είναι τα κατεπήγοντα θέματα τα οποία μένει να αξιολογήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την αξιολόγηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Πολιτικής Ασφαλείας στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε γύρω από τα θέματα αυτά τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΧΟΜ. Suite la directrice de μετά είναι και επίσης και η αναπληρώτρια διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης. Τους καλωσορίζω και τους δύο. Σας προτείνω την εξή μέθοδο. Μετά από τις παρουσιάσεις τους και μετά από την πρώτη παρουσίαση από πλευράς του κ. Νίδη, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, μια σειρά αν θέλετε ερωτήσεων, και μετά μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων και μετά τη δεύτερη ομιλία, μέσα σε μια μισή ώρα αυτά, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορέσουν να εκφραστούν και να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Συνεπώς λοιπόν σας ζητώ να μην καθυστερήσουμε άλλο, ο κύριος λοιπόν ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μπορείτε να μείνετε στη θέση σας είτε να έρθετε εδώ όπως θέλετε. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η πρώτη επίσκεψη την οποία κάνω στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και εξ ονόματος του Επιτρόπου Κίνγκ να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Είναι μια ειδική επιτροπή αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι σημαντικό, αξίζει τουλάχιστον μια τέτοια επιτροπή και είναι σαφές ότι και τα δικά σας φώτα και απόψεις θα είναι χρήσιμα για να προσανατολίσουμε καλύτερα τις εργασίες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας ευχαριστήσω επίσης που αυτή η δεύτερη συνεδρίασή σας αφιερώνεται στην αξιολόγηση η οποία μόλις ολοκληρώθηκε μάλλον τον μήνα Ιούλιο ολοκληρώθηκε, αξιολόγηση η οποία θα σας επιτρέψει νομίζω να έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήρη κατάλογο του τι έχει ήδη γίνει και γίνεται στον τομέα της ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα της τρομοκρατίας. Το κείμενο λοιπόν που έχω προετοιμάσει είναι στην αγγλική και γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσω στην αγγλική και θα παρουσιάσω και κάποιες διαφάνειες. Λοιπόν, οι τρεις παραδοσιακοί πυλώνες της πολιτικής ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Καταρχάς, είναι μια ανάλυση αυτή που κάναμε η οποία γίνεται στο εσωτερικό των υπηρεσιών μετά από ευρύτατες διαβουλεύσεις σε πολλές χώρες μέλη και σε πολλές υπηρεσίες και διεθνείς οργανώσεις και εμπλεκόμενα μέρη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα αποτελέσματα ο Επίτροπος Κίνγκ είχε την δυνατότητα να τα παρουσιάσει με συντομία στην Επιτροπή ΛΥΠ τα αποτελέσματα είναι θετικά. Απαιτούνται νέες, νέες δράσεις, είναι οι δράσεις αυτές που πρέπει να είναι φυσικά σχετικές και αποτελεσματικές. Βέβαια δεν είναι όλα τέλεια, δεν μπορούμε εδώ να καθησυχάσουμε, να εφησυχάσουμε ε, τις προσπάθειές μας, πρέπει να τις συνεχίσουμε και σε άλλους τομείς, τομείς στους οποίους μάλιστα η δική σας κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να είναι ιδιαίτερος υποβοηθητική, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε και να βελτιώσουμε τα μέτρα αυτά, έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, πρώτον, βλέπουμε ότι υπάρχει ατελής εφαρμογή εδώ είναι ένας τομέας στον οποίο οι δικές σας εργασίες ελπίζω να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε την όθηση που απαιτείται και να αυξήσουμε την πίεση και νομοθετικά και εκτός νομοθετικής ε, πλευράς, καλύτερη τεκμηρίωση σε τομείς όπως το PNR, τα προσωπικά στοιχεία επιβατών, η λειτουργική χρήση του συστήματος του Ευρωπαϊκού ξεκινάει από το Μάιο του 2018. Πολλές χώρες μέλη έχουν καθυστερήσει και υπάρχουν και άλλοι τομείς οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται συστηματικά στο κέντρο των συζητήσεων. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα νομοθετικά πλαίσια εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες πρακτικές δυσκολίες εφαρμοστικού τύπου. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η ενδογενής περιπλοκότητα του συστήματος και των διαφορετικών μέσων τα οποία έχουμε αναπτύξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βασική μας προτεραιότητα είναι να προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια να αναπτύξουμε κάποιους τομείς για καλύτερη συνεργασία να απλοποιήσουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας, το REFIT σαν παράδειγμα, να συμπληρώσουμε τις κατευθύνσεις και την καθοδήγηση εφαρμογή σαν παράδειγμα του κώδικα Schengen, του συνοριακού κώδικα στον τομέα των εκρηκτικών σαν παράδειγμα. Υπάρχει επίσης ένα άλλο θέμα, είναι η έλλειψη δυνατοτήτων των κρατών μελών. Υπάρχει έλλειψη πόρων, διότι υπάρχει ακριβώς τεράστια ζήτηση ειδικού τύπου υπηρεσιών. Αυτό το αισθανόμεθα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ισχύει για πόρους γενικότερα, αλλά και για εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επίπεδου στον τεχνολογικό τομέα, όπως την κρυπτογράφηση. Και τέταρτο βασικό συμπέρασμα είναι η ανάγκη ε, προσαρμοστικότητας, να είμαστε πολλαπλής χρήσεως, όχι μόνο να συνειδητοποιούμε την φύση του κινδύνου, αλλά ο τρόπος δράσης των τρομοκρατών εξελίσσεται, αλλάζει και γι' αυτό θα πρέπει να αποδείξουμε ότι τα μέσα μας είναι ικανά να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες αλλαγές. Για το ξεκινήσαμε κάπως να συζητάμε τα θέματα αυτά με διαφθρωμένο τρόπο κατά πολέμησης της τρομοκρατίας δηλαδή από το 2005 και μετά έχουμε προτείνει και αυτό επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο και το ε, Κοινοβούλιο μια κοινή στρατηγική. Οι ε, βασικοί κανόνες της στρατηγικής αυτής παραμένουν θα πρέπει να προσπαθήσουμε κάθε φορά να καλύψουμε όλες τις πλευρές και στον τομέα της πρόληψης, της προστασίας, της συνέχισης και της ανταπόκρισης στις απειλές και τους κινδύνους. Αυτή, αν θέλετε, αυτό το πλαίσιο αντιλήψεων, το βασικό πλαίσιο, εκπληρούνται σταδιακά. Πιστεύουμε ότι οι πιο πρόσφατες και χρήσιμες οριζόντιες μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η πρόσφατη οδηγία η οποία εξυγχρονίστηκε και έγινε δεκτή το Φεβρουάριο του 2017. Εμείς στα πλαίσια αυτής της νομοθετικής ρύθμισης θεωρούμε ότι οι συνομοθέτες στάθηκαν ικανοί να καλύψουν όλες τις πλευρές καταπολέμησης της τρομοκρατίας από το βασικό επίπεδο, το επίπεδο ορισμού, το τι είναι τρομοκρατία, μέχρι επίσης και τις διαδικασίες ποινικοποίηση όλων αυτών των δράσεων και κωδικοποίηση όλων των καινοτόμων τρόπων συνεργασίας από το απλό επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών μέχρι το περίπλοκο επίπεδο της επιχειρησιακής ανταπόκρισης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις ε, εμπεριέχουν και το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτο κομμάτι της θεματολογίας που θέλω να θέσω είναι θα έλεγα το βασικό πρόβλημα της ριζιστο, ριζοσπαστικοποίησης. Είναι κάτι το οποίο είδαμε πολύ έντονα σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει ένα μοναδικό τρόπο λειτουργίας, έχει ακολουθήσει μια πολιτική αντιριζοσπαστικοποίησης, έχει διαθέσει πιστώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο κέντρο και δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται από 2.400 επαγγελματίες οι οποίοι είναι παρόντες έτσι ώστε να παρέχουν τις απόψεις τους και τις οδηγίες τους για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πολύ περίπλοκο και σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Και οι δύο πλευρές πρώτον, δηλαδή ο εντοπισμός, η ανείχνευση των ριζοσπαστικοποιημένων προσώπων, βλέπουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αρκετά θετικά αποτελέσματα και η δεύτερη πλευρά εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και περισσότερη προσοχή. Είναι η λεγόμενη απόριζοσπαστικοποίηση. Και εδώ βλέπουμε ότι τελικά είναι σχετικά εύκολο να ανοιχνεύσουμε τα άτομα αυτά και να μπορέσουμε να απομονώσουμε τμήματα του πληθυσμού από την ριζοσπαστικοποίηση. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε τις σωστές προτάσεις για την λεγόμενη απορριζοσπαστικοποίηση των ατόμων αυτών. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα στον τομέα αυτό και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε και μια ομάδα υψηλού επίπεδου κατά τη ριζοσπαστικοποίηση. Είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένας από τους πολλούς παρατηρητές και εξετάζει η ομάδα αυτή νέους τρόπους, όχι μόνο για να θέσει εν παραλίλω τις εθνικές αρχές, και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους και την ποιότητα της ανταπόκρισης, της απάντησής τους, αλλά μια ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία θα εξετάσει και νέες θεματολογίες, δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο καλοί για την κάλυψη των αναγκών των πληθυσμών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως τα παιδιά και οι γυναίκες πώς θα μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι σε ειδικά περιβάλλοντα όπως το κατασταλτικό και το περιβάλλον το σοφρονιστικό, της φυλακές. Πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, φαινόμενα ε, ο ιδεολογικού τύπου και πώς επίσης θα μπορέσουμε να συμμαχίσουμε με χώρες γύρω από την Ευρώπη που έχουν εμπειρίες στον τομέα της απορριζοσπαστικοποίησης να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρία των Δυτικών Βαλκανίων. Χώρες από την περιοχή αυτή έχουν μεγάλες ανάγκες, όπως και στο βόρειο τμήμα της Αφρικανικής Υπήρου. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο έχουμε δει ότι συνεισφέρει στη ριζοσπαστικοποίηση των ευάλωτων πληθυσμών, το διαδίκτυο. Το είδος του περιεχομένου το οποίο διακινείται στο διαδίκτυο. Οι διαφορετικές μορφές του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να, να κηρύσσονται ιδεολογίες που οδηγούν στην ιδεολογικοποίηση της πίστης και την ριζοσπαστικοποίηση. Και εδώ προσπαθούμε να στραφούμε στην επίτευξη γρήγορα αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και σε συνεργασία με τους ε, εμπλεκομένους ε, στο ίντερνετ. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, έχει υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και τη επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμένη παρέμβαση στο διαδίκτυο. να υπάρξουν αναχώματα, δηλαδή στη διάδοση ε, του μίσους που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και που οδηγεί στην τρομοκρατία. Ε, έχουμε μεθόδους έτσι ώστε τα υλικά τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα να αποσύρονται Έχουμε αυτή τη στιγμή 160 κέντρα τα οποία συνεργάζονται για την απόσυρση περιεχομένου που θεωρείται επικίνδυνο, αλλά εκεί όπου ελείπει συνεργασία είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο διαδίκτυο, οι παράγοντες του διαδικτύου οι οποίοι θα πρέπει να εντοπίζουν μόνοι τους, να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι λοιπόν το υλικό αυτή στιγμή ανοιχνευθεί να μην είναι πλέον επισκέψιμο στα πλαίσια του διαδικτύου με οδήποτε τρόπο. Υπάρχουν ευρύτατα πεδία λοιπόν συνεργασία στον τομέα αυτό. Προσπαθούμε να βρούμε και διαφορετικούς τρόπους προστασίας αν θέλετε. Οι αρχικές προσπάθειες εδώ και 10 περίπου χρόνια έχουν συγκεντρώσει την προστοχή τους στην προστασία των λεγόμενων κρίσιμων υποδομών καθοριστικών υποδομών. Ήδη οι πρώτες προτάσεις ήλθαν το 2008. Η αξιολόγηση δεν είναι καλή για την οδηγία που εφαρμόζεται μέχρι τώρα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες γιατί η εμβέλεια της οδηγίας είναι πολύ περιορισμένη. Η οδηγία καλύπτει μόνο τις μεταφορές και την ενέργεια. Και ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την κάλυψη και διασφάλιση των δραστηριοτήτων αυτών είναι πάρα πολύ επιβαρημένος. Ο τύπος των υποδομών, καταγραφής των υποδομών ε, και η μέθοδος που ακολουθείτε δεν δίδει τα απαιτούμενε εγγυήσει, τα απαιτούμενα εχέγγυα για γρήγορη απάντηση, ανταπόκριση ε, των αναγκών όταν αυτές αποκαλύπτονται. Βασικός νέος στόχος είναι ο λεγόμενος ο δημόσιος χώρος. Είδαμε στις τελευταίες επιθέσεις ότι σε δημόσιους χώρους οι επιθέσεις αυτές εκτιλήσονται. Εδώ ο Επίτροπος Κίνγκ στην Επιτροπή Λίμπε ε, είπε ότι στις 18 Οκτωβρίου την Τετάρτη δηλαδή θα ανακοινωθεί μια πρώτη πολιτική για την προστασία των δημόσιων χώρων. Είναι θα έλεγα ένα βασικό βήμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο σωστά και να βοηθήσουμε όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τους δημόσιους χώρους έτσι ώστε ε, να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Τα μέσα τα οποία έχουμε από την φάση της αξιολόγησης του κινδύνου, του εντοπισμού των χώρων και των τρόπων παρέμβασης για, την, ε, ε, για να καταστούν οι χώροι αυτοί ασφαλέστεροι, εκμεταλλευόμεθα τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε ας πούμε σε ορισμένες διαδικασίες vetting, μιλάμε για δημόσιους χώρους, οπότε έχουμε να κάνουμε εδώ με πολλαπλής μορφής εταίρους, εντελώς διαφορετικής φύσεως. Οπότε θα πρέπει και οι οικονομικοί παράγοντες, σαν παράδειγμα, να συμμετέχουν. Επιχειρήσεις, σαν παράδειγμα θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια πρακτικά βήματα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χώρους αυτούς να μπορέσουν να ελέγξουν μόνοι τους κάποιες πιθανές μορφές απειλής. Ο σχεδιασμός των δημοσίων αυτών χώρων όπου συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος και επίσης η συνειδητοποίηση από πλευράς του κοινού των κινδύνων που μπορεί να δημιουργούνται στους χώρους αυτούς και να μπορούν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας άλλος παραδοσιακός τομέας τον οποίο έχουμε εξετάσει <clears throat> σε σχέση με τις κρίσιμες υποδομές όπως είπα και μετά από τις 11 ε, Σεπτεμβρίου είναι η χρήση του πυρηνικού κινδύνου, η πυρηνική απειλή, η ραδιολογική απειλή και η χημική απειλή. Από το 2010 και μετά έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο, το CBRN, σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και οι ιδιώτες εταίρους και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε πρώτα καλύτερα τους κινδύνους Δεύτερο, να φέρουμε σε επαφή τους εμπλεκομένους έτσι ώστε ε, να εντοπίζονται καλύτερα πάλι οι κίνδυνοι και να υπάρχει ενιαία χρήση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα, αυτός είναι παραδοσιακός μας στόχος, να προσπαθήσουμε δηλαδή να εφεύρουμε λύσεις έτσι ώστε να απομακρύνουμε εκρηκτικά, χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά στοιχεία απειλής και να βελτιώσουμε την κατάσταση εντατικοποιώντας τις πολλαπλές μορφές συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκομένους και όταν λέω εμπλεκομένους εννοώ τους παραγωγούς των υπηρεσιών προστασίας αλλά και τους χρήστες και παραγωγούς των προϊόντων αυτών όπως τα χημικά και τα πυρηνικά. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει λόγω της φύσης των επιθέσεων που έχουμε υποστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται στην αγορά όπλων, ατομικών όπλων και εκρηκτικών. Η νομοθεσία στα εκρηκτικά είναι θα έλεγα αρκετά παλαιά, εδώ και 7 χρόνια υιοθετήθηκε. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε ε, το τι απαιτείται για να δημιουργηθούν, να παραχθούν εκρηκτικές ουσίες και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βελτιώσουμε επίσης και το θέμα της δημοσιοποίησης επικίνδυνων συναλλαγών δηλαδή αγορές προϊόντων που μπορεί να δημιουργήσουν ε, ε, συνθήκες για παραγωγή εκρηκτικών. Καλή συνεργασία λοιπόν ανάμεσα στις αρχές ελέγχου και εποπτείας, αλλά και συνεργασία των οικονομικών παραγόντων των επιχειρήσεων. Εδώ απαιτείται συνεργασία μαζί τους, απαιτείται ε, βελτίωση των γνώσεων που έχουμε σχετικά με τον ρόλο και την θέση των υλικών αυτών και πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε ακόμα περισσότερο το τι είναι βελτιώσιμο και να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα και των δικών σας εργασιών έτσι ώστε να εμφυσίσουμε νέες ιδέες στην αξιολόγηση την οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Μια φιλόδοξη αξιολόγηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την αγορά αυτή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή εκρηκτικών. Στα ατομικά όπλα. Εδώ έχουμε εξυγχρονισμένα νομοθετικά μέτρα πρόσφατα στις αρχές του 17. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε μετά από τα τελευταία νομοθετικά μέτρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά, έχουν δημιουργηθεί εθνικά contact points, έχουμε κυκλοφορήσει πολλές μορφές στήριξης του μηχανισμού ελέγχου των ατοπικών όπλων of uh, uh, Συνεπώς λοιπόν έτσι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε σε μια δεύτερη φάση καλύτερα αυτούς οι οποίοι πολλούν τα ατομικά όπλα αυτά και τους τρόπους με τους οποίους κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ή να μην είναι εφικτό. Η χρηματοδότηση τώρα των τρομοκρατικών οργανώσεων. Εδώ έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε μέχρι τώρα το λεγόμενο τρίγωνο πρόληψη, διερεύνηση, απόκριση. Στον τομέα της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Για να το πετύχουμε αυτό, συγκεντρώσαμε την προσοχή μας στις πιο σημαντικές και πιο παραδοσιακές μορφές ε, ε, οικονομικών συναλλαγών, μεταφοράς πιστώσεων δηλαδή, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τρομοκρατικές ενέργειες. Βλέπουμε όμως ότι όλο και περισσότερο τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν μη συμβατικούς τρόπους <clears throat> οικονομικής υποστήριξης, μη συμβατικούς τρόπους πρόκλησης και συλλογής χρημάτων προστήριξη των δραστηριοτήτων τους. Οπότε πρέπει να αλλάξουν και από πλευράς μας οι τρόποι ανταπόκρισης. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν ε, τον ρόλο των διερευνητικών ομάδων που έχουμε, των ανακριτικών ομάδων και να είμαστε πιο ικανοί στον εντοπισμό του είδους των συναλλαγών, οι οποίες πιθανώς να χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες είναι πολλαπλών φύσεων. Τώρα, ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι ένας τομέας στον οποίο αναμένουμε πάρα πολλά από πλευρά σας νέοι προσανατολισμοί και νέες μορφές στήριξη από πλευρά σας πάντα. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι ένας νέος τομέας, είναι ένας τομέας ο οποίος μας απασχολεί από την αρχή της αναδίπλωσης, αν θέλετε, των προσπαθειών μας για την προστασία μας, αλλά στον τομέα αυτό πολλές βελτιώσεις απαιτούνται να γίνουν ακόμα. Ο πρώτος χώρος τον οποίο θα έλεγα τον έχουμε λίγο ξεχάσει όταν μιλάμε για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι η αξιολόγηση κινδύνου ασφαλείας. Εδώ έχει αποδειχθεί πλέον ότι συνολικά στα πλαίσια των κατασταλτικών δραστηριοτήτων. Είμαστε σε θέση, σε επίπεδο τακτικής αντίδρασης, να προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ελέγξουμε όχι μόνο τη φύση του κινδύνου, αλλά να μπορέσουμε να κατανείμουμε τα επίπεδα κινδύνου και να καθοδηγήσουμε έτσι την καταλληλότερη μορφή απόκρισης. Ένας άλλος τομέας στον οποίο θέλουμε να απαντήσουμε περισσότερο έχουν υπάρξει θα έλεγα μέχρι τώρα πολύ σημαντικά βήματα προοδού στον τομέα της προστασίας συνόρων όταν αποφασίσατε εσείς να δώσετε νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή στα πλαίσια των, της ανάλυσης που έγινε για τις ευάλωτες πλευρές της δραστηριότητάς της. Απαιτείται λοιπόν να ελέγχουμε σωστά όχι μόνο το επίπεδο κινδύνου αλλά και τις δυνατότητες απόκρισης που έχουμε. Στα πλαίσια της ανάπτυξης τώρα περαιτέρω των δυνατοτήτων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε εδώ έχουμε τη, ένα παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε χτίσει τόσο χρόνια. Πρόκειται για την Europol που έχει αυτό το κέντρο τρομοκρατικής δράσης. Οπότε εκεί Why? Because uh, the... θα, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί, διότι αυτή η υπηρεσία έχει μπορέσει να πλασαριστεί ως ε, το κατεξοχήν σταυροδρόμι και κόμβος όσον αφορά τις ε, πληροφορίες για όλη την Ευρώπη και σήμερα ε, έχει χειρισμό σε πάνω από 9.000 δραστηριότητες τρομοκρατικές και 30.000 ε, περιπτώσεις προειδοποιήσεων για κάποιους επισημασμένους Ευρωπαίους που έχουν ταξιδέψει σε περιοχές συγκρούσεων. Οπότε όλα αυτά θεσπίστηκαν και συγκροτήθηκαν στην Ευρώπη και όλα αυτά είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα στα κράτη-μέλη. Και όλοι επίσης παίρνουν το φορείο σε αυτές οι υπηρεσίες από το δίκτυο ΣΥΕΝ, αυτό το οποίο το έφτιαξε η Europol. Και αυτό το αντιτρομοκρατικό κέντρο, η CTC, με τα χρόνια αναπτύχθηκε έχει προσφέρει και εμπειρογνωμοσύνη ειδική φύσεως. Σήμερα δε ε, επιλαμβάνεται οποτεδήποτε έχουμε κάποια τρομοκρατική επίθεση σε κάποιο κράτος μέλος. Αυτό το κράτος μέλος και κοινοποιεί, έρχεται σε επαφή και ζητεί την βοήθεια του αντιτρομοκρατικού κέντρου. Και έτσι υπάρχει υποστήριξη σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, αλλά και εξοπλισμό Άρα θα μπει στο παιχνίδι η Ιντερπολ με πιο αναβαθμισμένο ρόλο στα πλαίσια του νέου κανισμού που θα διέπει τη λειτουργία και είπαμε ότι είναι πρόσφατος αυτός ο κανονισμός και θα συζήτησαμε την περασμένη εβδομάδα στην ενακτήρια σας συνεδρίαση και έχουμε αυτό το καινούργιο υποπτικό σώμα της, ε, για τη Europol ε, το κοινοβουλευτικό όργανο εποπτείας και, και έτσι θα εξασφαλίσουμε να έχει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες η Europol και κυρίως αυτό αφορά πληροφορίες από χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε από όλο τον κόσμο, οπότε έτσι θα αναπαθμιστεί ο ρόλος της Europol. Έτσι θα μας προσδώσει μια προσθεμένη αξία στη δράση δηλαδή των εθνικών υπηρεσιών και έτσι να έχουμε πιο ποιοτικέ πληροφορίες από πολλές χώρες, όσες προτίθενται να συνεργαστούν. Ε, άρα, βέβαια, χρειάζονται κάποιες ε, συμφωνίες, οι κατάλληλες συμφωνίες και γι' αυτό σύντομα θα δοθεί η έντολη για διαπραγματεύσεις με αυτές τις χώρες με τις οποίες εργαζόμαστε. The uh, uh, uh, έχουμε και τα συστήματα πληροφοριών. Ε, αφορούν τους τομείς όπου έχουμε επί εννέα μήνες αφιερώσει πόρους. Πολύ σημαντικός τομέας. Υπάρχουν τέτοια συστήματα πληροφοριών αξιόλογα, σφαιρικά, στην αλλά αυτά έχουν αναπτυχθεί μέσα στον χρόνο. Αυτά που λέμε διαλειτουργικά Έχουμε επομένω αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και όλες, όλους τους, τους ευρωπαϊκούς παράγοντες και εμπλεκόμενους, θεσμικά όργανα κλπ. Ούτω ώστε να γίνονται τα εξή σε τρει άξονε. Πρώτα από όλα να αξιοποιούμε καλύτερα τα υπάρχοντα συστήματα. Δεν θέλουμε να βρούμε νέα συστήματα σαν αυτό σκοπό. Όμω, όταν υπάρχει κάποιο περίπλοκο σύστημα όπω το πριν έχουμε κάτι το οποίο έχει περισσότερο διακυβερνητική φύση. Και έχουμε και άλλα συστήματα όπως το PNR για τους επιβάτες των επιβατικών αεροπλάνων και θέλουμε όλα αυτά να ωφελούν και σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το έχετε συζητήσει πολλές φορές επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι να βελτιωθεί και η προσβασιμότητα και το τι είδος πληροφοριών θα καλύπτονται όπως το, σύστημα του Σέγγεν, του Eurodac και τελευταία το ECRIS. Θα σας τα πει τώρα η συνάδελφος. Δεύτερος άξονας, να μπορούμε να άρουμε κάποια κενά τα οποία υπάρχουν για κάποια συστήματα που δεν υπάρχουν, να βρούμε κάποια συστήματα που χρειάζονται και έτσι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις δυνατότητες του να επισημένονται οι ενδυνάμοι δράστες για προμονητικές απόπειρες. Και στο ΕΤΙΑΣ επίσης θα συμπληρώνεται ε, αυτό, αυτό το σύνολο συστημάτων πληροφοριών. Άρα να αξιοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα τα υπάρχοντα συστήματα. Άρα εντίθεση από την αμερικανική προσέγγιση κατόπιν των επιθέσεων της 10 Σεπτεμβρίου δεν θέλουμε να είναι κάτι κατευθυνόμενο. δεν θέλουμε να έχουμε ένα κεντρικό πρωτόκολλο αρχείο μητρό πληροφοριών. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα συστήματα ούτω ώστε να τα υποστηρίξουμε, να κάνουμε έλεγχο της ποιότητας των πληροφοριών, ότι μπαίνει στα υπάρχοντα συστήματα να υπάρχει μια μηχανή αναζήτησης, να μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα αυτούς τους πιθανούς ε, υπόπτους, πιθανούς δράστες και τα βιομετρικά να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Διότι έγινε στις πρόσφατες ε, επιθέσεις πάρα πολλές φορές. Κάποιοι κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στη ζώνη Σέγγεν με διαφορετικές ταυτότητες, αλλά πρώτη προτεραιότητα είναι να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών, να εξασφαλίσουμε το ότι κάποιος δεν θα μπορεί να αποκτήσει νομότυπα διαφορετικές ταυτότητες και να αξιοποιήσουμε το βιομετρικό υλικό που έχουμε. Τέλος. Όσο αφορά την επιχειρησιακή υποστήριξη που υπάρχει σε επίπεδο ένωσης, να σταθώ σε ό,τι γίνεται στις διάφορες υπηρεσίες. Αυτές που έχουμε συγκροτήσει και εξελίξει μέσα στα χρόνια το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ήταν υπέρ της εξέλιξης αυτών των υπηρεσιών. Και άρα θα πρέπει το μήνυμα να είναι το ότι χρειάζονται περισσότερες υπηρεσίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες. Εκτιμούνται πάρα πολύ από τις εθνικές αρχές και από άλλους ομολόγους ας πούμε στις χώρες που συνεργαζόμαστε. Άρα θέλουμε περισσότερους πόρους, περισσότερη γνωμοσύνη για αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε κατακλείδη το μήνυμα, το συμπέρασμα της αξιολόγησης ποιο είναι. Πρώτα πρώτα, πλήρης εφαρμογή και υλοποίηση. PNR, εκρηκτικά, όπλα. Πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη στήριξη και βοήθεια σε αρχές για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα εργαλεία που τους έχουν διατεθεί. Οι περιπλοκόντες τώρα των σχετικών εργαλείων. Εδώ είναι ευθύνη μας το να τα απλουστεύσουμε, να τα κάνουμε καταλληλότερα για τους σημερινούς στόχους. Ε, αυτό και γίνεται όσον αφορά και τις πληροφορίες στα συστήματα δεδομένων. Να ανταποκρίνονται, να αντιδρούν ούτως υπήν καλύτερα αυτά τα συστήματα Τώρα για δημιουργία δυνατοτήτων δεν είναι μόνο αυτές οι υπηρεσίες, αλλά είναι και το ότι υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη υποστήριξη στα ευρωπαϊκά δίκτυα, ε, φέρει πίν το δίκτυο κατά της ριζοφραστικοποίησης, το RAN, ή επίσης και το δίκτυο Atlas. Και αυτό είναι κάτι που είναι τώρα πρωτοφανέ, δεν υπήρχε. Και έτσι οι εθνικέ αρχέ καταπολούν την δημοκρατία και αποφάσισαν με την υποστήριξη τη Ένωση να συγκροτήσουν ένα τέτοιο δίκτυο το οποίο να λειτουργεί ούτω ώστε να βοηθάει τον κράτο στο άλλο και επίσης να μπορεί να επανέλθει σε περίπτωση επίθεσης και να παρεμβαίνει δηλαδή υπέρ του πληγέντος κράτους μέλους. Τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποια ευελιξία γιατί πάντα θα πρέπει να μπορούμε να αντιδράσουμε ή στις αλλαγές για το μόντους operandi των τρομοκρατών. στο δημοσιο χώρο, στον κυβερνοχώρο γιατί δεν το είπα προηγουμένω, αλλά και εδώ όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιείται ο κυβερνοχώρο από του ε, τρομοκράτε. για να κρυφτούν, για να μπορέσουν να κάνουν τι επιθέσει του και για την ριζοπραστικοποίηση. Αυτό είναι νέο, αλλά είναι και κάτι που επήγει για όλε τι αρχέ. Άρα θα πρέπει να είμαστε θέση να βοηθήσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Και Τώρα έχει την σκητάλη η Ευχαριστώ πρόεδρε. Πραγματικά πολύ καλή η δουλειά και η παρουσίαση. Έχετε λάβει είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή. Σας υπενθυμίζω το πολύ καλό αυτό έγγραφο που θα συμπληρωθεί από το έγγραφο της 18 Οκτωβρίου που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ εξ ονόματι όλων των συναδέλφων για την παρουσίαση αυτή που σίγουρα θα έχει δημιουργήσει απορίες και ερωτήματα. Η ε, κυρία Τίνα Άστολα, αν κατάλαβα καλά, ήθελε και αυτή τώρα να πάρει το λόγο και μετά θα συλλέξουμε τις ερωτήσεις και θα περάσουμε στο γύρο των απαντήσεων. Αλλά θα σας παρακαλέσω να μην μακρηγορήσετε όσο ο προλαλής σας συνάδελφό σας για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να έχουμε ένα γύρο ερώτα απαντήσεων αξιότιμοι βουλευτέ και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να έρθω εδώ για να σας παρουσιάσω τα μέτρα που αντιλαμβάνει η ΓΔ δικαιοσύνη στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η εντολή της επιτροπή σας ε, δείχνει πολύ ξεκάθαρα ότι οι πολιτικές για την ε, μείωση των τρομοκρατικών απειλών είναι πολύ σημαντικές οι επιθέσεις ήταν απρόβλεπτες ε, και το είδαμε και τελευταία. Μεγάλη πρόκληση για τις δημοκρατίες ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απειλές ε, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τις αξίες της Ευρώπης. Η ασφάλεια λοιπόν αλλά και η ελευθερία είναι συμπληρωματικές, αλληλοενισχυόμενες αενίες και στόχοι της πολιτικής που χαράσει και η στρατηγική η δική μας γενική διεύθυνση θα σας πω ποιες αρχές έχει. Πρώτα απ' όλα, καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να έχουν ε, τα μέσα στη διάθεσή τους για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και επίσης θα πρέπει να αποτραπεί η ριζοσπαστικοποίηση, το ανέφερε και ο προλαλής σας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο μας για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης ε, τις πηγές δηλαδή που χρησιμοποιούν τρομοκρατές και εγκληματίες, πώς μπορούμε να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Είχαμε την οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος ε, πρόσφατα. Τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί πράγματι στη επιτόπου από όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε λοιπόν προς το παρόν να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Και η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας έχει ξεκινήσει και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή πολιτική. Προς τον τομέα αυτό Περιβαίνοντας ε, και τις, ε, το, το εντολή της Διεθνούς ε, Task Force για τον τομέα αυτό, ελπίζουμε ότι μπορεί να εξευρεθεί το του δυνατό πολιτική απόφαση. Ο συνάδελφός μου προανέφερε τις μονάδες πληροφοριών στον τομέα της χρηματοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν αυτές τις μονάδες πληροφοριών και να υιοθετήσουν ένα συντονισμένο σύστημα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία την περαιτέρω και να τους παράσχουμε ενισχυμένες εξουσίες. Οι δικαστικές αρχές τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μια κοινωνία που δέπεται από το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντική στο ρόλο της Eurojust για την ε, διευκόλυνση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικές υποθέσεις. Τα κράτη-μέλη αναζητούν την ε, βοήθεια, τη συνδρομή της Eurojust στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο και από ό,τι γνωρίζω έχουμε 69 έρευνες αυτή τη στιγμή ε, για θέματα τρομοκρατίας. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούγκερ, θέλουμε να δούμε και κατά πόσον ε, το EPPO, δηλαδή ε, το γραφείο του Σαγγελέα, θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες ε, με προοπτική το, και χρονικό ρίζο το 2025. Σίγουρα το γραφείο του Σαγγελέα πάρα πολύ αποτελεσματικό. Εμείς θέλουμε να είναι πιο επιχειρησιακό και πιο αποτελεσματικό με μια αναθεώρηση των ε, δομών διακυβέρνησης και ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την πρόταση που καταθέσει Κομισιόν στο επίπεδο του τεμερούς διαλόγου. Από ό,τι γνωρίζω και εσείς ε, σχεδιάζετε επίσκεψη στη Eurojust τις ε, επόμενες εβδομάδες. Εκεί θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από κοντά τι δουλειά γίνεται. Η Eurojust έχει εντοπίσει σημαντικές προκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, τις διώξεις και γενικότερα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια δέσμη προκλήσεων, δηλαδή η συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων και των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόσβαση στις πληροφορίες ε, και από ένα λογαριασμό email, από το υπολογιστικό νέφος κτλ καθιστούν πιο δύσκολο το έργο των διοκτικών αρχών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται συχνά σε ξένες χώρες και γι' αυτό εργαζόμαστε να βρούμε τα πρακτικά μέτρα για να βοηθήσουμε τους ε, εισαγγελείς και τους υπεύθυνου ε, των διοκτικών υπηρεσιών για να ε, αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας του χρόνου θα παρουσιάσουμε μάλιστα νομοθετική πρόταση για την διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι κάτι που ήδη αναφέρθηκε και το κεντρικό σύστημα που επεξεργαζόμαστε, το ECRIS, TCN, θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε και πληροφορίες για καταδίκες ε, υπηκών τρίτων χωρών. Ελπίζω να συνεργαστούμε πολύ καλά και να έχουμε και επιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων το συντομότερο δυνατό. Τη διαλειτουργικότητα την ανέφερε ο συνάδελφος σε σχέση με τις, ε, πώς να το πω, με αυτά τα σιλό πληροφοριών και βέβαια τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να υλοποιήσουμε αυτή τη διαλειτουργικότητα αλλά επαγγελματάς πλήρως ε, για τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον 21ο αιώνα πραγματικά είναι εφικτό και να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας ακόμη περισσότερο. Με δημιουργία έξυπνων λύσεων θα περιλαμβάνουν ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων και έχουμε και τις ε, σχετικές ε, οδηγίες που είναι πολύ σημαντικές. Πέραν τώρα των δεδομένων προσωπικού ναι. χαρακτήρα, τα μέτρα ασφαλεία θα πρέπει να συνάδουν με τι αρχέ τη αναγκαιότητα και τη αναλογικότητα, όπω προβλέπει ο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Προ τούτο λοιπόν εξετάζουμε όλε τι προτάσει για να δούμε τι αντίκτυπο θα έχουν για τα δικαιώματα αυτά και θέλουμε να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τα κράτη-μέλη, να σέβονται ταυτόχρονα όμως και τον χάρτο των δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έχουμε τη νέα οδηγία για την καταλλήλωση των επικρατές που ενέκριναν φέτος Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Είναι ένα καλό παράδειγμα των κοινών προσπαθειών. Ελήφθησαν ήδη λοιπόν υπόψη ορισμένε πτυχέ που έχουν να κάνουν με το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα στη διαδικασία τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση. Οι αρχέ αναγκαιότητα και τη αναλογικότητα μεταξύ ή το δικαίωμα έκφρασης, ελευθερίας διακίνησης. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Στην οδηγία αυτή υπάρχει σαφής ρήτρα για τα θεμελιώδη δικαιώματα για πρώτη φορά. Και γίνεται λόγος για εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτού του εργαλείου για να δούμε ποιο θα είναι ο αντίκτυπο τη ελευθερία ελευθερίες και δικαιώματα. Τώρα, λίγα λόγια για την πρόληψη ή αποτροπή της ε, ριζοσπαστικοποίηση και του εξτρεμισμού. Με μια κοινωνία με αλληλεγγύη, χωρίς αποκλεισμού και πιο ε, με μεγαλύτερη ε, ανθεκτικότητα. Θέλουμε να αποτρέψουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, να καταπολεμήσουμε τη μυσαλλοδοξία και την ρητορική μίσους. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε τη στιγματοποίηση, το στιγματισμό ομάδων ή κοινοτήτων που μπορεί να απολώσει τις κοινωνίες. Οι εκφάνσεις ε, ε, ε, είναι η ε, ρητορική μίσους όπως είπα, μυσαλλοδοξία κτλ. Έχουμε το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβία. Συμφωνήσαμε να έχουμε κώδικα συμπεριφορά για τις μεγαλύτερε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, για την καταπολέμηση της ε, ε, σε πράξεις μίσους, όπως αυτή γίνεται μέσω διαδικτύου. Και πράγματι αυτές ε, οι ομιλίες ή αυτές οι τα μηνύματα μίσους ε, πλέον διαγράφονται πάρα πολύ γρήγορα από το διαδίκτυο. Το τελευταίο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και μια ανακοίνωση για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου, του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου με μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, αρχών για την αναβάθμιση του παράνομου περιεχομένου από τις διάφορες πλατφόρμες και συνεργασία με κράτη-μέλη, αρχές και άλλους φορείς. στη ριζοσπαστικοποίηση τώρα στις φυλακές. Θέλω να αναφερθώ. Θέλουμε να επιτρέψουμε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να βοηθήσουμε στη χρηματοδότηση. Το Φεβρουάριο του χρόνου θα οργανώσουμε ένα συνέδριο με δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλους οπλιστικών καταστημάτων για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ένα σημαντικό στοιχείο που ίσως είναι και μια αφετηρία, είναι εναλλακτικές ε, μορφές αντί της κράτησης, ιδίως για τα παιδιά και τις γυναίκες. Ίσως καλό θα ήταν ολοκληρώσω εδώ. Θέλω να πω ότι περιμένω με υπομονησία το feedback για τις προτάσεις επιτροπής σας ελπίζοντας να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας και οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά σε μια ανοιχτή κοινωνία χωρίς περιορισμούς. Σας ευχαριστούμε κυρία Άστολα για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ και γιατί σεβαστήκατε το χρόνο αγόρευσης. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Θα πρότεινα καταρχάς το λόγο να έχουν οι συντονιστές εφόσον τον επιθυμούν, να τον λάβουν και μετά ε, όποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να, να μιλήσουν. Η κυρία Αναγκόμες είναι η πρώτη βουλευτής που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Θα ήθελα την αξιολόγηση, την εκτίμησή σας για αυτά τα σιλό που είπατε. Μήπως αυτή ε, η στεγανοποίηση κατά κάποιο τρόπο μας επηρεάζει αρνητικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και έχω για μια ερώτηση. Έχετε εκτιμήσει τις δυνατότητες ή την έλλειψη δυνατοτήτων των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το νομικό και συνταγματικό τους πλαίσιο για τη διεξαγωγή βασικών επιχειρήσεων και δράσεων. Πάντα βέβαια σύμφωνα με το δίκαιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σε θέματα αναχέτηση ανταλλαγή πληροφοριών κτλ. κτλ. Γιατί αν δεν γίνεται νόμο και γίνεται παράνομα, έρχεται μπούμεραγκ σε ό,τι αφορά την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης. Ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθείτε για την ε, αντιμετώπιση, την απόρριψη και την εναλλακτική λύση σε εισαγωγή ημάμιδων από χώρες όπως το Πακιστάν για παράδειγμα. Αν αυτό ε, το κάνετε με προβλεκτικό, με proactive τρόπο. και αν υπάρχει και κάποια συνεργασία με τέτοιες χώρες. Επίσης, PNR, τα στοιχεία επιβατών. Δεν είναι πανάκια, δεν εφαρμόζεται, αλλά τέλος πάντων. Από την αρχή υπήρχε ένα πρόβλημα για το ότι δεν καλύπτεται τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Ιδιωτικά αεροσκάφη λοιπόν τα οποία προσγειώνονται σε ενωσιακά αεροδρόμια δεν θα πρέπει να ερευνώνται. Πώς θα το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να φέρουν και ταγκόν και ε, ε, ναρκωτικά, οι οικογένειες ολόκληρες ε, μέσα. Πώς θα ελέγχονται, θα έπρεπε να ελέγχονται. Και τέλος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εδώ έγινε και το ερώτημά μου. Ε, τα συλλόγια γιατί δεν καταλαβαίνω. Έχω συμμετάσχει στη χάραξη της ομοθεσίας για την καξάπλημα χρήματος. Ήδη από την πρώτη οδηγία και μέχρι την τέταρτη. Και βλέπω ότι καθυστέρουν, κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις λύσεις. Και στο πλαίσιο της πέμπτης οδηγίας ενώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. αποσιάζει όμως πλήρως από όλη τη συλλογιστική. Πώς θα προχωρήσουμε, διαρωτώ με. Είμαστε σοβαροί ή δεν είμαστε. Η Κομισιόν πρόσφατα, διαστόματος Μοσκοβισή, ή των υπηρεσιών του Μοσκοβισή τέλος πάντων, είπε ότι το σύστημα ΦΠΑ το εκμεταλλεύονται για τη χρηματοδότηση των νομοκρατών. Μιλάμε για τεράστια ποσά. πέντε δι το χρόνο. Δεν μιλάμε για προπληρωμένε κάρτες. Δεν έγινε λόγο γι' αυτό. Γάμα Δέλτα Τάξου, Γάμα Δέλτα Γιούρι δεν συνεργάζονται στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα που βλέπουμε να εκμεταλλεύονται τις, τις λειτουργίες μας στο φορολογικό επίπεδο οι τρομοκράτες. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Merci, euh, Anna Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Άντερς Φίστηγεν, που είναι ο συντονιστής για το ECR. Παρακαλώ να είστε συντομότεροι τόσο ώστε να μπορέσουν να λάβουν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι. Και μετά ο Ζων Φιλίπ Άλμπρεχτ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δευτερολογήσει. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να προσπαθήσω να συμμορφωθώ με αυτό το χρονικό όριο που τώρα επιβάλλεται. Α δούμε για πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ σφαιρική, συνολική, πλήρη για τα συμπεράσματά μα χρήσιμη και θέλω να σταθώ σε κάποια θέματα όπου θέλω να μου τα εξηγήσετε λίγο περισσότερο πρώτα πρώτα όσον αφορά τις συστάσεις στη σελίδα 81 λέτε εκεί στη σύσταση λέει 8 ότι τα ευρωπαϊκά όργανα και η Διευθυντική Επιτροπή Εταιρεών θα πρέπει πιο δυναμικά να εμπλακεί ε, ούτως ώστε να υπάρχει αυτού του είδους το πουλ των εμπειρογνωμόνων αλλά και εκπροσώπων ε, του κλάδου. Εδώ θέλουμε ότι τα εργαλεία που ήδη έχουμε θα πρέπει να αξιοποιούνται περισσότερο και ε, θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να μην ε, θεσπίζουμε καινούργια πλαίσια και καινούργια εργαλεία. Οπότε πέστε μου την άποψή σας. Πώς με τον καλύτερο τρόπο στο μέλλον θα μπορέσουμε να, το κάνουμε αυτό και από την αρχή να, είναι πιο πλήρες η δράση μας και να μην προσπαθούμε να παρέχουμε για να φτιάξουν τα κοσκήμενα εκ των υστέρων σαν το PNR, ε, το Schengen, το σύστημα και τα σύνορα. Πώς τα βλέπετε. Α, α τελειώνει όμως το δίρετο, οπότε να σας πω το ότι βέβαια έχουμε για τις εσωτερικές πολιτικές αυτή τη μελέτη, αλλά έχετε εξετάσει το τι γίνεται από πολλές εξωτερικές πολιτικές. Μας είπατε κάτι για τη Μέση Ανατολή, μας είπατε για τις χώρες από Αφρική και από Ασία. Ασχοληθήκατε καθόλου προς τα εκεί και να συνδέσετε και αυτή τη δουλειά προς τα έξω με αυτό που γίνεται εντός Ένωσης. Προσπάθησα, Πρόεδρε, να τηρήσω το δίλεπτο, αλλά ελπίζω να με συμπαθήσετε, να με συμπαθάτε, να με συγχωρήσετε τέλος πάντων για την υπέρβαση. Ναι, ευχαριστώ συνάδελφε που τηρήσατε το δίλεπτο και τώρα. Άλμπρεχτ. Και εσείς δύο λεπτά. Και εδώ πριν έχουμε την πρώτη σειρά απαντήσεων για αυτές τις ερωτήσεις. Άλμπρεχτ. ευχαριστώ πρόεδρε. Για πέστε μας. Τι γίνεται και με κάποιες άλλες μέλες που υπάρχουν από ειδικού για αυτά τα θέματα, μια που η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται την τελευταία δεκαετία, μην πω δεκαπενταετία, είναι πολύ σημαντική. Και όλο ένα και πιο φανερό καθίσταται ότι θα πρέπει εμείς να συζητήσουμε πώς οι διοικητικές αρχές θα εφαρμόζουν όλα αυτά τα οποία έχουμε θεσπίσει. Αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε, όχι να βρίσκουμε καινούργια, καινούρια μέτρα. Άρα αυτό να προσέξετε. Και έχουμε πει και την πρικοδότηση κάποιων κοινών ερευνητικών ομάδων καλύτερη συνεργασία διοικητικών αρχών, δικαστικών αρχών και έτσι θα χρησιμοποιούνται τα ισχύοντα μέτρα. Γιατί υπάρχουν μελέτε εξόλου που λένε πάρα πολλά από αυτά τα μέτρα στι τελευταίε 15 ετία ελήφθησαν, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Υπήρχε κάποιο στρατηγικό πλάνο και επειδή κάτι έπρεπε να γίνει για να αντιδράσουμε κατά κάποιο τρόπο, τα θεσπίσαμε, αλλά πώ γίνεται να μου καλύτερε επιδόσει στο μέλλον στρατηγική, ε, μελέτες επιπτώσεων, να έχουμε αυτές τις ρήτρες βαθμιάς κατάργηση. αυτές τις sunset clause τέλο πάντων και αναθυδά. Το, το μελετάτε το ω μια επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Και τώρα να δώσουμε τον λόγο πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσουν σε αυτή την πρώτη σειρά ερωτήσεων. Yes, uh, maybe I take... Ε, κάπως αντίστροφη σειρά να ακολουθήσω η τελευταία ερώτηση ότι έχουν πάρα πολλά μέτρα, δεν έχουμε μελέτες επιπτώσεων. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ε, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε μέσα από τις κρίσεις. Και αυτού του είδους η συνολική αξιολόγηση έγινε για να μπορέσουμε να έχουμε μια γενική έποψη του πώς έχει το τοπίο, πώς έχουν τα πράγματα. Και σωστά είπατε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την αξιολόγηση των εργαλείων. Να έχουμε αυτές τις ρήτρες για τα εργαλεία να βελτιώνουμε τα υπάρχοντα εργαλεία. Είναι βασικό αυτό. Αυτά προσπαθούμε τώρα να περιχαρακώσουμε για αυτήν την αξιολόγηση. Τώρα όσον αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων και αυτό εύστοχο που είπατε. Είπαμε ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση για πάρα πολλά εργαλεία ακόμα ισχύει η περιπλοκότητα των εκτήρων της εφαρμογής. Επομένως, όποτε κάνουμε κάποια αναθεώρηση, είτε της νομοθεσίας, είτε του ορισμού, είτε ακόμα και της προοικοδότησης, να προσέχουμε να μην περιπλέκονται τόσο πολύ τα πράγματα για αυτό που θέλουμε να βοηθήσουμε. Κάθε φορά. Άρα, απλούστευση. Άρα, προτάσεις για κάποια πράγματα που πρέπει να είναι πιο εύληπτα, πιο κατανοητά. που αποτριότητα είναι όχι να έχουμε και άλλη νομοθεσία σε οποιοδήποτε τομέα, εκτός από το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αυτό το οποίο είπαμε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά που τα έχουμε επισημάνει. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αντί για την νομοθεσία να έχουμε υλικό, να έχουμε κατευθυντήριε γραμμές ας πούμε. Κάτι άλλο επίση το οποίο είπαμε είναι το θέμα της ε, ε, εκπαίδευσης, κατάρτισης. Έχουμε αυτή την ΣΕΠΟΛ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε για την εκπαίδευση των ε, διοικητικών αρχών των διαφόρων υπηρεσιών να την αξιοποιήσουμε την ΣΕΠΟΛ να τους δώσουν περισσότερους πόρους. Τώρα αφορά την εξωτερική πτυχή, τις εξωτερικές σχέσεις ας πούμε, είναι θέμα οριζόντιο σε αυτή την αξιολόγηση και η βασική προστιθέμενη αξία πρώτα πρώτα είναι το θέμα των κυρώσεων πολύ σημαντικό άλλο σημαντικό παραδοσιακά είναι το πραγματικό δίκτυο που διαθέτει η Ένωση και επίσης το τι γίνεται με τους αντιτρομονετικούς διαλόγους που έχουμε αναπτύξει διαχρονικά σχεδόν με όλες τις χώρες που μπορούν κάπως να συμβάλλουν που έχουν κάνει τέλο πάντων οι ίδιες κάτι στον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Να τι μας λέει η υπηρεσία δράσεις δράσης και άλλοι φορείς της πολιτικής. Τώρα, πώς μπορούμε σε επίπεδο πολιτικής να ωφεληθούμε από τους ασχολούμενους στην πράξη με αυτά. Είναι σωστό, θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα και εκεί, καλά λέτε. Το είπαμε και αυτό στην ε, αξιολόγηση, να προσέξουμε τι λένε αυτοί που ασχολούν στην πράξη, που εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα. Και θα πούμε για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορίας και πληροφόρηση είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εμπλέξουμε όλους τους εμπειρογνώμους. Ε, γι' αυτό και τελικά έχουμε πιο αποτελέσματα, που είναι επικοδομητική αυτή η προσπάθεια να, όπως τώρα κάνουμε και με αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Έχει υπάρξει συζήτηση κατόπιν προτάσεις και έτσι να ξέρουμε τι χρειάζεται από αυτού που στην πράξη ασχολούνται με αυτό τώρα όσον αφορά το συλλογικό. Και εδώ θα γίνει αξιολόγηση και εδώ περιμένουμε τη συμβολή. Υπάρχει μια προστορία 15 ετών σε αυτό το μέτωπο και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Έχει υπάρξει πολύ καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ε, αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Ας πούμε, οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών έχουν καλύτερα συνεργαστεί. Τα τελωνία, το ίδιο. Η συνοριοφυλακή σε κάθε κράτος. Μας θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Ακριβώς αυτό έχει επισημανθεί σε κάθε κράτος που προσπαθεί κάτι να κάνει για την τρομοκρατία. Να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις αρμόδιες αρχέ. Και γι' αυτό που είπατε για τη χρηματοδότηση. τα τελωνία. Ακόμα και οι φορολογικές αρχές έχουν κάποιες μεθοδολογίες. Υπάρχει μέθοδοι αξιολόγηση κινδύνου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις παραδοσιακές διοικητικές αρχές. Και ο Επίτροπος Κίνγκ αυτά θέλει να κάνει σε επίπεδο ασφάλειας. Να συγκεράσει τις διάφορες επιμέρους δραστηριότητες. να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά μέσα. Α, όπως ο κ. Μασκοβίση λέει για την ε, φορολογία. Έτσι δηλαδή, να μπορούν να δρουν καλύτερα οι ίδιες Πολύ σημαντικά αυτά. Τώρα, όσον αφορά αυτού του είδους την δυναμική προσέγγιση για την καταβολή της ριζοσπαστικοποίησης, μας αναφέρονται δύο παραδείγματα γιατί τη χρηματοδότηση σε κάποιες χώρες για κάποια μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εθνικέ αρχέ. και έτσι να φροντίσουμε για την κοινωνική δράση κάποιων θρησκευτικών κέντρων. Λεπτό το θέμα. Υπήρξε όμως ε, συνένεση ε, εκεί στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και να τα κοιτάξουμε έτσι αυτά γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες, κατανόηση του προβλήματος και να μπορέσουμε να βρούμε τις απαντήσεις στα διάφορα θέματα με περισσότερη διαφάνεια για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποιος κώδικας διοντολογίας, σωστής πρακτικής ας πούμε και να υπάρχει κάποιο είδου ευρωπαϊκή συμφωνία. Πού να θεσπίζει κάποιες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτω ώστε να διαχειριστούμε αυτά τα ζητήματα. Α, ακριβώς όπως κάνουν οι αρχές για διάφορους οργανισμούς τώρα. Για το PNR φυσικά και δεν καλύπτει τα ιδιωτικά αεροσκάφια υπάρχουν κενά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε. Οι εθνικές αρχές προσπαθούν να ασχοληθούν περισσότερο, γιατί ας πούμε οι εθνικέ αρχές όταν υπάρχει χρήση ιδιωτικού αεροσκάφου κοιτούν τι είδου ε, άδεια ε, πτήσης κυκλοφορία υπάρχει. όμως εδώ δεν είμαστε πάντοτε εναρμονισμένοι. Ε, Γι' αυτό και χρειάζεται η ανάλυση κίνδυνου. Ποτέ δεν θα υπάρχουν όλα τα μέσα, τα εργαλεία, ούτω ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος κάθε εισόδου, κάθε μεταφοράς, κάθε μέσο μεταφορικού. του όμως να μοιράζονται τις πληροφορίες, να κάνουν την ανάλυση του κινδύνου με καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά το πώς θα κάνουμε τη διαφορά. Τι Τι κάνουν τα κράτη-μέλη και τι δεν κάνουν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δική μας δουλειά να πάμε σε ένα κράτος μέλος και να κάνουμε κάτι. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες να δώσουμε μέσα εργαλεία στα κράτη-μέλη πρέπει να το διαπραγματευτούμε αυτό καλά μαζί για να τους καλύψουμε τις ανάγκες. Το θέμα της βυσοσπαστικοποίησης της φυλακές είναι ναι, θα έλεγα ένα θέμα σημαντικό και εδώ οι ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα στις διάφορες χώρες πολύτιμες. με το νέο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας όταν συμπεριληφθεί πλέον στις αρμοδιότητες του EPPO τα πράγματα θα είναι πιο ελεγχόμενα. Το θέμα της εφαρμογής, της σταδιακής εφαρμογής, αυτό είναι το θέμα που τίθεται μόνιμα σε σχέση με την εφαρμογή του κοινοτικού νόμου. Υπάρχουν ε, διαδικασίες σεμιναρίων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επίσης χρηματοδοτούμε και τη Eurojust ε, η οποία έχει και τις μικτές ανακριτικές ομάδες που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις επακριβέστατες απαντήσεις σας που δημιουργούν και άλλα ερωτήματα βέβαια. Δίνω το λόγο στη Μαϊτέ για δύο λεπτά, η οποία αντικαθιστά το Ζεράρντε Πρέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ίσως να τις έχετε εξηγήσει επανειλημμένα, αλλά εγώ ομολογώ εδώ τα κενά τα οποία έχω σε σχέση αυτό. Το πρώτο αναφέρεται στα θέματα της εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής οδηγίας έχει περάσει, θα έχει περάσει ε, τον Σεπτέμβριο του 18 ένας χρόνος περίπου από τώρα. Σε ποια φάση πιστεύετε ότι θα έχουμε φτάσει και πώς θα γνωρίζουμε αν πράγματι σε όλες τις χώρες αν εφαρμόζεται ή σωστά αυτό το οποίο προβλέπει σε ποιοτικό επίπεδο η οδηγία. Δεύτερον, στις 3 Ιουλίου του 17 έγινε μια μεγάλη κλοπή σε στρατιωτική μονάδα της ε, Πορτογαλίας ε, και κλάπησε μια ολόκληρη σειρά πολεμικού υλικού, χειροβομβίδες, αυτόματα. Εκλάπη επίσης και μια, ένα φορτηγάκι με στρατιωτικό υλικό, εν πάση περιπτώσει. Όλες αυτές είναι κρίσιμες υποδομές επικίνδυνες για τις κρίσιμες υποδομές και έχει υπάρξει θα έλεγα κάποια συνεργασία. Έχετε πληροφορίες γύρω από τα δύο αυτά συμβάντα γιατί τα θέματα αυτά για το επίπεδο ασφαλείας μας ενδιαφέρει είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ κύριος Βανόρντεν, Δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Βανόρντεν. Διερωτώ αν μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εδώ μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και μια αξιολόγηση ειδικά των αντιτρομοκρατικών πολιτικών. Το θέμα είναι ότι τα έγγραφα αυτά που παράγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσει να παράγει δυστυχώς λίγοι τα διαβάζουν. Διερωτώ με λοιπόν πού θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τελικά την προσοχή μας. Η δική μου άποψη είναι να μην αναζητήσουμε επιπλέον ρόλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ίσως να υπάρχει κάποιος ρόλος εφόσον δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Στα πλαίσια των παρατηρήσεών μου λοιπόν, πού θα πρέπει να βάλουμε την προτεραιότητα. Θέλουμε να επισκεφθούμε τη Europol, τη Eurojust και τη Frontex σε κάποια φάση. Μπορούμε να πάμε εκεί, να μείνουμε ώρες, να μας ενημερώσουν. Αυτό όμως τώρα δεν μας δείχνει το πού θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ συνάδελφε για δύο λεπτά. Ο κύριος Οτζούλητσα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε κάποιο γραπτό υλικό και στα έγγραφα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά θεωρητικά στοιχεία και λίγα πολύ πρακτικά στοιχεία. Είναι απρόβλεπτες ε, οι τρομοκρατικές ανάγκες. Αν πράγματι υπήρχε η απαραίτητη συνεργασία ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας, ε, τις δυνάμεις συλλογής πληροφοριών κτλ. νομίζω ότι θα ήταν λιγότερες οι επιθέσεις αυτές. Το να παράγεται ένα επιπλέον έγγραφο χωρίς καμία μεγάλη σημασία δεν μας βοηθάει. Λέει εδώ ποιες είναι οι αδυναμίες του συστήματος, τι δεν δουλεύει σε εθνικό επίπεδο, τι δεν δουλεύει σε κοινοτικό επίπεδο, γιατί αλλιώς τα έγγραφα αυτά θα είναι κενό γράμμα. Σήμερα το απόγευμα είχα πάει στο Κυργιστάν. Ένα από τα θέματα ήταν οι ξένοι μαχητές. Υπάρχουν όλοι και περισσότεροι από αυτούς τους ξένους μαχητές του ΝΤΑΕΣ που ητάτε αυτή την εποχή που θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση λοιπόν και αυτού του φαινομένου και όχι μόνο σε γενικόλογο επίπεδο. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές βοήθειας στον κόσμο, το 50%, 56% προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω της βοήθειας αυτής τα προγράμματα για την απορριζοσπαστικοποίηση. Πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε σωστά τους ξένους μαχητές οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα για να μην είναι πλέον ριζοσπαστικοποιημένοι. Ε, χώρες όπως η Βοσνία, Ευζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Αλβανία. Υπάρχουν εκατοντάδες μαχητές από τη Συρία που επιστρέφουν εκεί. Τι γίνεται με τις χώρες επίσης της Βόρειας Αφρικής που παίρνουν βοήθεια από μας. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε μέσω των χρημάτων που δίδουμε για βοήθεια να βοηθηθούμε και εμείς για την εφαρμογή των μέτρων αυτών που μας αφορούν. δυστυχώς το τμήμα καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Αεροπόλ δεν είναι λειτουργικό ουσιαστικά, απλά συλλέγει πληροφορίες. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Χρειάζεται σωστή συνεργασία ανάμεσα στις διοκτικές αρχές και σωστή συνεργασία ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Πολιτική συνεργασία δηλαδή. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν τεράστιοι αριθμοί τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχει η απαιτούμενη συνεργασία. Αγαπητέ συνάδελφοι, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. Για να μπουν και οι υπόλοιποι να πάρουν το λόγο και να κάνουν τι ερωτήσει του. Μίλαν Σβέρ, ο επόμενο. Και Αρνό Ντανζάν. Μόλι ζήτησε το λόγο που τη βλέπω. Α, ξέχασα την Κατερίνα Κινίτσι. Άρα η Κατερίνα Κινίτσι πρώτα, μετά ο Μίλαν Σβέρ και μετά ο Αρνό Ντανζάν και εδώ κλείνει ο κατάλογος και ακολουθούν οι Απαντής. Κατερίνα, δύο λεπτά σας παρακαλώ. Εσείς ελπίζω να σεβαστείτε το χρόνο σας, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις με αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι κανένα πρόβλημα. Τι απλώς ξέχασα. Ε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα τόσο ενδελεχή τα οποία μας εξήγησαν για την αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών πολιτικών. Είναι πολύ περίπλοκη η υπόθεση και χαίρομαι που αναφέρθηκε η οδηγία που ελήφθη υπόψη αυτή η προσπάθεια συγκερασμού ασφάλειας με τα κριτήρια της αναλογικότητας και σεβασμού των δικαιωμάτων. Όλα αυτά θα χρειαστεί αυθεντική πρόληψη η οδηγία όπως και άλλα πρόσφατα νομοθετήματα εξυγχρόνισαν τα εργαλεία τα αντιτρομοκρατικά. Όμως πια αυτά δεν αρκούν. χρειάζεται συνέχεια να λαμβάνουμε υπόψη πώς εξελίσσεται η τρομοκρατία. Πρώτα πρώτα σίγουρα χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών. Η ε, ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων για την χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας, άρα χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης θέμα της κρυπτογράφησης, κωδικοποίησης και αυτό θα είναι θέμα που θα έχουμε αύριο και το θέμα των αποδεικτικών στοιχείων. Στη Europol ε, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά σε πολλά κράτη όχι. Άρα εδώ πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση και πώς επομένως θα είναι σημείο να σε γύρω πολλά από τα κράτη-μέλη. Να κάνετε μια αξιολόγηση πάνω σε αυτό. Για τα αποδεικτικά στοιχεία τώρα. Για τι ηλεκτρονικές, ηλεκτρονικό χαρακτήρα αποδείξει. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούν οι, οι έρευνες, να γίνει εδώ αξιολόγηση, θα έχουμε κάποια πρόταση σύντομα. Έχει γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων έχει γίνει προκαταρκτική μελέτη με συγκεκριμένο χαρακτήρα. Τι γίνεται για τις δέουσες μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας. Ε, μα είναι πάρα πολύ μπερδεμένο το θέμα. Άρα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας σε βάθος. Ευχαριστώ κύριο Σβέ για δύο λεπτά. Επαναλαμβάνω την επιθυμία μου να μπορέσουμε να ακούσουμε όλους. Άρα να σεβαστείτε παρακαλώ το δίλεπτο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις παρουσίασεις, την παρουσίαση αυτής της πάρα πολύ καλής ε, έκθεσης. Είναι καλά και αποτελεσματικά όπως φαίνονται, αλλά νομίζω ότι είναι και υπεραισιόδοξα. Διότι από τη μελέτη νομίζω ότι το αντίθετο προκύπτει ως συμπέρασμα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποια συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο κρατών μέλων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει επίσης επαρκή συνεργασία ενώ στη ΣΥΠΑ φαίνεται το πρόβλημα να έχει αντιμετωπιστεί. Δεν έχω πολύ χρόνο για να επεκταθώ. Αναφέρθηκε το πολύ σημαντικό πρόβλημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί στην προσέγγιση τους. Σε ό,τι δεν αφορά το ομοθετικό πλαίσιο έχουμε τα μέσα, αλλά διερωτώμε με πώς γίνεται το Ιρανικό καθεστώς μέσω του τραπεζικού συστήματος και μέσω μιας σλοβενικής τράπεζας ε, σε μια χώρα να έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει το ένα δις για τη χρηματοδότηση, ένα δις μάλλον για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού του προγράμματος. Οι αστυνομικές αρχές θα πρέπει να ερευνήσουν ε, πάρα πολύ ε, την κατάσταση. Υπάρχει και μία περίπτωση ενός εμβάσμου 80 εκατομμυρίων ε, στην Γερμανία. Η Επιτροπή Πάναμα για τα Panama Papers επίσης πρέπει να κάνει και αυτή την δουλειά που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τώρα ο Αρνό Ντανζά και μετά η κυρία Στίβενς με την οποία θα κλείσει ο κατάλογος. Κύριος Ντανζά, δεν είχα αποφασίσει να πάρω το λόγο, αλλά θέλω να αντιδράσω σε αυτά που ακούω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κοτολογίες και μεγάλα λόγια να λέμε εκτός πραγματικότητας. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται κάτι. Είπατε για την Πορτογαλία που υπήρξε αυτή η κλοπή μεγαλύτερη. Κάποιος είπε στρατητικού υλικού. Όχι. Φυσικά και έχουν υπάρξει πολύ μεγαλύτερε πριν από δύο χρόνια, στη Γαλλία για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό τη Πορτογαλία. Άρα να μένουμε στα γεγονότα, τα πραγματικά και να λέμε πιο μεγάλη κλοπή έγινε κτλ. Για του ξένου μαχητέ ε, επιστρέφουν μαζικά, ακούγεται. Μα δεν, ε, δεν ισχύει. Πριν από κάποιου μήνε γύριζαν πολύ περισσότεροι από ότι τώρα. Μπορεί να ανατραστραφεί αυτή η τάση και να επανέλθουν περισσότεροι. Προ το παρόν όμω δεν γίνεται αυτό. Δεν επιστρέφουν μαζικά. Για τον πολύ εντό αγωγικών καλό λόγο ότι σκοτώνονται στα πεδία της μάχης ε, εκεί. Και γι' αυτό γυρίζουν λιγότεροι πίσω. Τώρα, για τη συνεργασία. Μην λέμε ότι όλες οι επιθέσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έγιναν γιατί δεν υπήρχε συνεργασία. Υπήρξαν πάρα πολλές επιθέσεις οι οποίες αποσοβήθηκαν γιατί υπήρχε καλή συνεργασία και το θέμα είναι να δούμε και ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες. Γιατί δεν μπόρεσαν αυτές οι επιθέσεις που πέτυχαν να είχαν αποσοβηθεί. Υπάρχουν επιθέσεις στην Ισπανία, ε, στην ε, ε, Γαλλία και σε άλλες χώρες που ε, έγιναν γιατί δεν μπόρεσαν να ε, έχουν εντοπιστεί οι δράστες νωρίτερα, γιατί ίσως δεν υπήρξε κατάλληλη συνεργασία των ε, δικτύων των διοκτικών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε, να δουλέψουμε σοβαρότητα, αλλά να δούμε πρώτα απ' όλα και τις πληροφορίες. Δεν τις έχουμε ακόμα όλες τις πληροφορίες και γι' αυτό δεν πρέπει να συνάγουμε βιαστικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ η Χέλγα Στίβενς τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, από τη Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Ονιντή για την παρουσίασή του και τις δύο παρουσιάσεις τις ε, μελέτησα και έχω και κάποιες ερωτήσεις για τις αυτές εκθέσεις. η ανάλυση καταρχάς ε, των ανοιχτών πηγών, open source. Είναι μια αναφορά στην ανάλυση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Αρμόδιο Κέντρο. Το σκανάσμα των email λοιπά. Υπάρχουν κάποια λογισμικά που μπορεί κανείς να τα βρει και στο διαδίκτυο και με αυτά μπορεί να βρίσκει λέξεις, μηνύματα που να παραπέμπουν σε τα κτλ. Το Βέλγιο στα τέλη της χρονιάς αγόρασε αυτό το υπερλογισμικό από τη διάβασα για να βοηθηθεί η Εθνική Υπηρεσία για να μπορεί να μπαίνει στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web και να ανακαλύπτει αυτά τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να αγοραστεί το λογισμικό αυτό ε, ή αν υποστηρίζονται τέλο πάντων τα κράτη-μέλη που θέλουν να αγοράσουν αυτό το λογισμικό από την και Ξέρετε κάτι για τέτοιου είδου ε, τεχνολογίες και δυνατότητες. Επίσης, μια κεντρική μονάδα που θα βοηθούσε τα ζητήματα κρυπτογράφησης. Ε, πώς το βλέπετε ως ιδέα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο. Εσείς δεν ήσασταν εγγεγραμμένος. Τέλος πάντων. Άντε, να σας δώσω ένα λεπτό. Αλλά όχι παραπάνω, γιατί είχα κλείσει τον κατάλογο. Κύριε ένα λεπτό. La parole à nous deux intervenants. Και μετά θα απαντήσουν ο κύριος Έλισεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο και την κυρία από την Κομισιόν για τις παρουσιάσεις τους. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ο κύριος Ονιντή μίλησε για την ιδεολογία και το ρόλο της και η κυρία Άστολα μίλησε για την πρόληψη αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης και ότι πρέπει να αντιδρούμε από τον προτέρων. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν έχετε ασχοληθεί και με κάτι άλλο. Το ρόλο και τις χρηματοδοτικές ροές από και προς τεμένη και υπάρχει κάποια παρακολούθηση, κάποιο έλεγχο των ριζοσπαστικοποιημένων ημάμιδων. Τι δυνατότητες υπάρχουν για έγκαιρη αντίδραση. Δηλαδή θα ήθελα λίγο να επεκταθείτε στο ρόλο της ιδεολογίας και τι γίνεται στα τεμένη ό,τι αφορά χρηματοδοτικές ροές. Για την ε, κήρυξη μίσους, για την ε, ρητορική μίσους που ασκείται εκεί. για το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας κατά πολέμησης τρομοκρατίας. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή τον πίνακα αποτελεσμάτων αναχώρα. Αλλά εμείς έχουμε τακτικές συναντήσεις με όλες τις χώρες της Ένωσης και δεν έχω μηνύματα ιδιαίτερων δυσκολιών. Αυτό που θα κάνω ίσως να σας δώσω γραπτά μια περιγραφή της κατάστασης. Κανία χώρα δεν έχει ανακοινώσει την πλήρη μεταφορά στην παρούσα φάση. Ελπίζω να σας στείλω πιο επακριβείς πληροφορίες τώρα για το ρόλο των ιδεολογιών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το οποίο εμείς αναζητήσαμε στα πλαίσια της συζήτησης ε, της ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης είναι ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι ήταν γενικά καλή ιδέα συλλογικά να υπάρξει μια επεξεργασία θέσεων κατανόησης της ιδεολογίας και των ιδεολογιών στην διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι ώστε με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, πανεπιστημιακών και ε, εργαζομένων στους τομείς αυτούς να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε καλύτερα και να καταπολεμήσουμε καλύτερα κάποιες οργανώσεις, να καταπολεμήσουμε την χρηματοδότησή τους και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ιδεολογία τους. για το ρόλο καλύτερης ανάγκης για καλύτερη συνεργασία. Να απευθύνω μια έκκληση και προς εσάς πριν απ' όλα να πω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να αναγνωρίσουμε ότι τα πράγματα σε ένα βαθμό λειτουργούν. Στα, ιδιαίτερα στα πλαίσια μια σημαντική συνεισφοράς και από τη δική σας Επιτροπή, να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους λοιπόν για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Να συνειδητοποιήσουμε την βάση από την οποία έκινησα. Όλες οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή λόγω της σημερινής κατάστασης λειτουργούν στο φουλ, κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να ε, επικοινωνήσουν καλύτερα και μεταξύ τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εσωτερικά σε κάθε χώρα ανάμεσα στις διαφορετικές αρχές και για να απαντήσω εδώ στον κύριο Βάνο Όρντεν. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα αν πραγματικά αφιερώνατε κάποιο από το χρόνο σας για να επισκεφθείτε τις τρεις οργανώσεις και να μπορέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και σε αυτές τις υπηρεσίες ε, να τους δώσετε την δυνατότητα να εκφραστούν, να ακούσετε αυτούς οι οποίοι καταπολεμούν την τρομοκρατία και να προσπαθήσετε να καταλάβετε καλύτερα τις ανάγκες τους έτσι ώστε όχι μόνο να μας διαφωτίσετε περισσότερο για το είδος των μέτρων τα οποία μπορούμε να προτείνουμε, αλλά και να μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βοηθώντας τις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταλάβουν καλύτερα όπως τα θέματα της πολιτικής, της εμπορικής, των χρηματαγορών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο πιο κατανοητό έτσι ώστε να δούμε τις αδυναμίες που έχει το σύστημά μας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Σχετικά τώρα με τα υπόλοιπα στα οποία αναφερθήκατε σήμερα, φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, ανάγκη να υπάρξει μια ανάλυση για την περαιτέρω διευκόλυνση της ροής πληροφοριών, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η συνεισφορά σας νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Τώρα για, τους, ε, αυτούς που επιστρέφουν τους μαχητές, τους ξένους μαχητές. Πολλά έχουν γίνει ε, και σε επίπεδο ένωσης για αυτούς που είναι γνωστό ότι μάχονται σε ξένα εδάφη. Υπάρχουν ε, βελτιώσεις, εδώ πολλές, ένα μικρό παράδειγμα, όταν επισκεφθείτε την Ευρωπόλ θα υπάρξει δυνατότητα για την Ευρωπόλ να παίξει πλήρως τον ρόλο της ως γέφυρας ανάμεσα στις πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τρίτες χώρες εταίρους και τις εθνικές αρχές έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στην Ευρωπόλ την ευθύνη να τροφοδοτήσει με στοιχεία τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Δεδομένων. Αυτού του είδους τα παραδείγματα νομίζω ότι θα ε, οδηγήσουν σε πρακτικές βελτιώσεις γύρω από την συλλογή όλων των μεμονωμένων στοιχείων των σχετικών με τους ξένους μαχητές σε διάφορους τομείς και δεύτερον θα δώσουν τις καλύτερες δυνατότητες στην παρούσα φάση συνεργασίας και μέσω της Ευρωπόλ αλλά και μέσω τρίτων χωρών εταίρων. Για το θέμα της κρυπτογράφησης είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, τομέας. Θα σας τα εξηγήσει συνάδελφο σε λίγο. Σε σχέση με τα τεχνικά και τεχνολογικά θέματα αποφασίσαμε και αυτό θα είναι τμήμα του πακέτου καταπολέμησης τρομοκρατίας την Τετάρτη να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο την Europol σαν πραγματικό κέντρο αριστείας αν θέλετε έτσι ώστε όλες οι χώρες μέλη να προσφεύγουν εκεί για την αποκρυπτογράφηση υλικού που κρύβεται συνήθως σε hardware το οποίο χρησιμοποιούν οι εγκληματίες και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνικών γνώσεων των εθνικών αρχών έτσι ώστε οι εθνικές αρχές να είναι πάντα πολύ προχωρημένες στα πλαίσια του ελέγχου των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες. Και τέλος, για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο και, τους, α, και τις αναλύσεις ανοιχτού κώδικα πηγής. Νομίζω ότι εδώ και στα πλαίσια των συζητήσεων με τις εταιρείες του διαδικτύου αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι ο κόσμος του διαδικτύου πρέπει να μας βοηθήσει να εντοπίζουμε στοιχεία υλικά και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτες ε, για να ριζοσπαστικοποιούν και ε, να προσλαμβάνουν σε εισαγωγικά ε, ανθρώπους για εξυπηρέτηση των στόχων τους. Θα πρέπει οι μηχανισμοί του ίντερνετ να χρησιμοποιήσουν κάποια μέσα παρακολούθησης στον τομέα φυσικά της τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να εντοπίζουν αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν τα στοιχεία αυτά. Υπάρχει ένα όριο για μας ε, το τι μπορούμε να ζητήσουμε από τις ε, επιχειρήσεις αυτές και η Europol και τα κράτη-μέλη, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε πάνω από το 15 με 20% των στοιχείων που κυκλοφορούν. Και γι' αυτό απαιτείται οι ίδιες οι επιχειρήσεις να κάνουν προσπάθεια και να δείξουν το ίδιο επίπεδο καινοτομία το οποίο επιδεικνύουν σε εμπορικό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει θα έλεγα και το δικό μας πρόγραμμα δράσης. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα τέθη, πού να εστιάσουμε Φοβούμαι ότι είναι ένας τομέας αυτός που χρειάζονται όλα τα διαφορετικά εργαλεία και πρέπει να ληφθούν υπόψη διαφορετικά βήματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να εστιάσουμε ή να επικεντρωθούμε κάπου, αλλά η πρόληψη σίγουρα είναι κάτι σημαντικό και είπα εναλλακτικέ επιλογές αντί της κράτησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πρόληψη έχει να κάνει και με την επιστροφή των ξένων μαχητών, χρηματοδότηση προγραμμάτων εξόδου, που τα λέμε, να μπορούν δηλαδή να βγουν από αυτό το ρόλο. Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε τα κράτη-μέλη προ αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και έχει υποθεί πολύ εδώ και θα το ξαναπώ εγώ να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτή. Θα γίνει μελέτη αντικτύπου στις αρχές του έτους. Ιδεολογία. Η ελευθερία έκφραση είναι κάτι πολύ σημαντικό και φυσικά και θέλουμε να παραμείνει. Στην Ευρώπη όμως υπάρχει ε, ποινικοποίηση της ε, ρητορικής μίσους ε, και γι' αυτό ε, μπορούμε να δράσουμε ε, στον τομέα αυτό και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος από τα απαντήσεων. Μπορεί να μην καλύφθηκαν οι συνάδελφοι, ήταν πολλές ερωτήσεις. Αν λοιπόν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να απευθύνετε γραπτό στους δύο προσκεκλημένους, μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω θέρμα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, για αυτό το διάλογο, που είναι και το πρώτο, ένα από τα πρώτα, αν θέλετε, λιθαράκια της Επιτροπής μας. Δηλαδή, να σε αυτό τη δυνατότητα να αποκτήσουμε κάποια γνώσεις, μία γνώση, όχι τέλεια γνώση ακόμη, αλλά τέλο πάντων να αρχίσουμε να έχουμε μία γνώση και ε, προσέγγιση για να προχωρήσουμε σε εργασίες μας. Με τους συντονιστές θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση με τις εργασίες μας θέλοντας να καλύψουμε όλες τις ε, εκφάνσεις. Θα είναι πολυδιάστατες οι συνεδριάσεις μας. Βέβαια, δεν θέλουμε να έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν θα το διαβάσει κανείς και δεν θα είναι και καθόλου χρήσιμο. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ούτε θέλουμε να κάνουμε τους ανήξερους ε, και ότι τώρα τα ανακαλύπτουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε απαντήσεις. Φυσικά και δεν αποκαλύπτονται όλες οι πληροφορίες, δεν ε, είναι γνωστό το έργο γενικώ και η αποσόβηση επιθέσεων ε, πάντοτε. Το θέμα λοιπόν είναι να έχουμε ενημέρωση, να έχουμε έναν απολογισμό. Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Και καλό να υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί. Που θα έρθει να προσθεθεί στη συνεργασία που υπάρχει ήδη μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών για να έχουμε πιο πολύ ε, συγκεκριμένες απαντήσεις ε, για τον πολίτη που περιμένει ακριβώς απαντήσεις από την Ευρώπη. Αυτή θα είναι και μια προκλήσεις μας, αναμφίβολα, να υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε πρακτικά εφαρμόσιμες προτάσεις και συστάσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ λοιπόν για μια ακόμη φορά. Θα έχουμε τη δυνατότητα εκ νέου να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ γιατί καταφέρατε να παρουσιάσετε συνθετικά το πολύπλοκο αυτό το οποίο και προσκαλώ εκ νέου τους συναδέλφους να έρθουν σε διμερή επαφή μαζί σας εφόσον θέλουν κάτι ακόμη να σας πούν. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης που είναι η παρουσίαση της μελέτης ε, από το θεματικό τμήμα δικαιωμάτων των πολιτών και των συνταγματικών υποθέσεων. Το θέμα της μελέτης είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τρεις είναι οι πτυχές, συνάφεια, συνοχή και αποτελεσματικότητα. Η κυρία Μπίμπη Βαν Γκίνκελ από το Διεθνές Κέντρο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας ACCT και ο κύριος Βιμ Βένσικ. Τον ξέρουμε καλά τον κύριο Βένσικ, γιατί ξανά ήταν εδώ. Από... από την Pricewaterhouse. Να σας ακούσουμε λοιπόν και αφού καλύψετε το θέμα σας. Ελπίζω σε 15 λεπτά θα έχουμε έναν γύρο ερώτα απαντήσεων. κύριε Βαν Δύσκολο να σας τα πω όλα αυτά σε ένα τεταρτάκι. Και συμπαθάτε με. Και το αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ παραγωγική ώρα που αυτό το μέτωπο είναι θέμα αποτελεσματικότητας και συντονισμού. αυτό θα σας πω. Είχαμε την έκθεση ε, της ε, Άνοιξης τον Ιανουάριο μετά και Φεβρουάριο του 2017, οπότε είχαμε ε, μετά κάποιες εξελίξεις αν μπορούμε να επικαιροποιήσουμε την έρευνα και οπότε με μεγάλη μας χάρη πιστώσαμε ότι κάποιες συστάσεις ελήφθησαν υπόψη και είναι σημαντικό αυτό για τους ερευνητάς. Ότι δηλαδή να πιάνουν τόπο αυτά που γράφουμε εμείς. Για να δούμε την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Στόχος της μελέτης. Κάνουμε μια καταγραφή του τι ισχύει σε αυτό το περιπλοκό θέμα, που έχουμε τόσους πολλούς εμπλεκομένους, οπότε και αυτό εξετάσαμε. τι έχει χρησιμοποιηθεί, τι πολιτικές υπάρχουν, πώς αλληλοσυνδέονται, αν υπάρχει κάποια νομιμοποίηση και συνάφεια αυτών. Τι έχει συμβεί. Μα τι να σας υπενθυμίσω. Ό,τι και να πω κάτι θα λείπει γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το επισημαίνουμε για να δούμε ότι τα πράγματα είναι σε συνεχή εξέλιξη και συνεχώς αναγύπτουν νέα. Έχουμε αυτούς τους μοναχικούς λύκους Θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Γιατί πια δεν χρησιμοποιούνται μόνο τα οχήματα, αλλά μαχαίρια κουζίνας. Άρα πώς να τα προλάβουμε. Υπάρχει εδώ θέμα του πώς θα υπάρξει μια προειδοποίηση. Και έχουμε εδώ και τους soft targets, τους πιο ανυπεράσπιτους ας πούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό, εάν τα δούμε τα πράγματα πιο μακρόπνο, να δούμε την εξέλιξη των τάσεων, θα καταλάβουμε καλύτερα το ότι έχουμε τώρα ποικιλία και όσον αφορά τους δράστες και όσον αφορά τους στόχους. Βλέπετε εδώ πως έχουμε αύξηση όσον αφορά αυτές τις επιθέσεις των μοναχικών λύκων, αλλά για τον αριθμό των επιθέσεων που κάνουν. Στην επόμενη διαφάνεια μιλούμε εδώ πέρα για αυτού του είδου την ε, ποικιλία, τη διαφοροποίηση στους στόχους. Πρώτα πρώτα ξεκινήσαμε με στόχους όπως στρατιωτικού στόχους, ε, ε, κρατικές υποδομές. Τώρα όμως βλέπουμε ποικιλία. Όλα μπορεί να είναι στόχος. Άρα θα πρέπει οι υπηρεσίες ασφαλείας εντοπίσουν ένα έργο ακόμα πιο δύσκολο. Θα πρέπει κανείς να προλάβει πολύ μεγαλύτερη βεντάλια από στόχους. Δεν έχουμε περιλάβει το, τι γίνεται ανά περιοχή, γιατί μιλήσαμε για αυτούς που γυρίζουν από τα πολεμικά μέτωπα, για τους ε, μαχητές επιστρέφουν οι ξένοι μαχητές. Οπότε και εδώ θα πρέπει να εξεταστεί τι διαφορές υπάρχουν, πού πάνε αυτοί. Και όπως είπατε χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Θα πρέπει να έχουμε ανάλυση από αυτόν των πληροφοριών, θα πρέπει να έχουμε προγνωστικά επί τη βάση ανάλυση των ιστορικών δεδομένων για να ξέρουμε τι μας έρχεται, τι θα μας συμβεί. Ε, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα τη λέει στον συνάδελφο. Για να δούμε τώρα, λέει ο κύριο. Ε, με την επόμενη διαφάνεια δούμε όλα αυτά τα προγράμματα, δράσεις στρατηγικές, συγκεκριμένα μέτρα βλέπουμε εδώ πέρα μια απότομη αύξηση μετά από κάποια επίθεση πολύ συχνά δεν έχουμε στρατηγική που για ένα μέτρο, αλλά μια τρομοκρατική επίθεση που το φέρνει. Για να δούμε τώρα όσα έχουν επιτευχθεί. Διαχρονικά σε πάρα πολλού τομεί, ακριβώ όπω τα εξήγησε προηγουμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ περιλαμβάνεται επίση και ένα μέτωπο το οποίο θεωρούσαμε ότι δεν είναι στην εντολή σα. Τα θέματα δηλαδή εκρηκτικών και όπλων. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό έχει συνάφεια με την εντολή σα, αλλά δεν καλύπτεται από την μελέτη μας. Θα μπορούσε όμως να περιληφθεί στο έργο της Επιτροπής σας κάτι. Νομίζω ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη, εάν ήδη δεν ανησυχούν, θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν για το ραδιόλο, και περισσότερες δυνατότητες δημιουργούνται από πλευράς των ε, τρομοκρατών. όλο ένα και καλύτερη γίνονται όσον αφορά την προπαγάνδα. Αλλά και όσον αφορά την τεχνολογία για τα χρηματοοικονομικά. Εάν σα ανησυχεί η χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, αρχίστε να ψάχνετε τι γίνεται με τα κρυπτογραφημένα νομίσματα, τι γίνεται με τους παρόχους υπηρεσιών χρηματοδότησης κλπ. Αυτά που δεν καλύπτονται σήμερα μέτρα. Οπότε εδώ επίσης έχουμε και τους soft targets και για σημαντικά έργα υποδομής. Πολύ σημαντικό σε αυτός ο τομέας θα πρέπει να καλυφθεί από τα μέτρα τα αντιτρομοκρατικά. Να την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ, αν δείτε τα της διαβίβασης δεδομένων, συνεργασία και ασφαλείας συνόρων έχουμε βήματα πρόοδου που έχουν επισημανθεί από την μελέτη μας για αυτό την, α, το να δίνει ένα τέλο πάντων τα δεδομένα στον άλλο. Αλλά πριν τη διαβίβαση και τη συνεργασία θα πρέπει να γίνει συλλογή δεδομένων ποιότητος. Άρα χρειάζονται σημαντικές αξιόλογες δυνατότητες επί το κράτους μέλους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. μπορούν όλοι να συλλέξουν ποιοτικά δεδομένα. Οπότε, ακόμα και με τις καλύτερες πλατφόρμες, πάντοτε κάτι θα πρέπει να μαζέψει κανείς. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντρογνωτικής Δραστηριότητα. και την πλατφόρμα που συνδυάζει πληροφορίες και δράση αλλά θα πρέπει να δούμε και πάλι τα της εντολής αυτών των υπηρεσιών και φυσικά πάντοτε υπάρχει ο συσχετισμός των δύο επιπέδων. Βέβαια κάθε κράτος μέλος του δομές καμιά φορά αυτό το κάνουν η αστυνομία, δηλαδή την αντιτρομοκρατική δραστηριότητα, καμιά φορά το έχει η υπηρεσία πληροφοριών ως έργο, καμιά φορά και οι δύο. Πολλές φορές έχουμε και άλλες υπηρεσίες φορολογικές, τελωνιακές Οπότε θα πρέπει να εξασφαλιστεί, του λαμβάνουμε υπόψη αυτής, αυτή την, την ποικιλία εθνικών δομών. Και έτσι εντελεί των πληροφοριών να βελτιωθεί. Όσον αφορά τη διαχείριση των σύνορων, διαπιστώσαμε ότι έχουμε ένα σωρό μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και κάποια συστήματα που έχουν προωθηθεί με χαρακτήρα αντιτρομοκρατικό. Το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εμεί. Το είπανε στη μελέτη αξιολόγηση όταν προσπάθησαν να διαπιστώσουν αν υπάρχει προστιθέμενη αξία για διάφορα είδη εγκληματικότητα, αν βοηθάται η ασφάλεια. Και είπαμε ότι για την αγώνα κατά της είναι περιορισμένη η προστιθέμενη αξία. Πολλέ φορές όμως προωθούνται αυτά τα συστήματα διαχείρισης συνόρων έτσι κι αλλιώς. Να ληφθεί αυτό υπόψη στην αξιολόγηση. Επόμενο. Όπως το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αντιμετώπιση όσον αφορά την διαβίβαση των πληροφοριών και αυτό αφορά και την ασφάλεια των συνόρων. Πάμε στο επόμενο. Τώρα για να δείτε εδώ πέρα τι όλες αυτές τις επιτροπές, όλους αυτούς που εμπλέκονται. Όπως είπατε, εδώ τα καταγράψαμε. Έχουμε εδώ πορτοκαλί, τη δική σας επιτροπή που είναι η πιο φρέσκια σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια επιτροπών. Βλέπετε ότι είναι δύσκολο κανείς να έχει μια άποψη για τι συμβαίνει για όλο το τοπίο και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός όλων αυτών σε επίπεδο συμβουλίου, σε επίπεδο ένωσης. Ε, υπάρχει αυτός ο συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης. Ε, το κάνει αυτό ο Επίτροπος Κίνγκ. Τώρα έχει ευρύτερη εντολή για να καλύψει και την τρομοκρατία. να δούμε επομένω όλα αυτά πώ συγκεράζονται, πώ συμπληρώνονται, να δούμε πώς θα υπάρχει η κατεύθυνση όλων προς την ίδια ρότα. Άρα, η επόμενη διαφάνεια, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς μπορεί να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε αυτούς τους τρεις άξονες, σε αυτές τις τρεις πολιτικές. Έχουμε κάποια συμπέρασματα, κάποιες συστάσει. Κάποιοι βουλευτές ήδη παρέπεμψαν στη δουλειά μας πριν. Ήδη υπάρχουν κάποια εργαλεία και άρα δεν είναι θέμα ε, επινόησης καινούριων εργαλείων, αλλά βελτίστων υπαρχόντων αλλιώ απλώς σωρεύονται περισσότερα. Θα πρέπει να ξέρουμε, να ξέρουμε ποιες είναι οι απειλές, θα πρέπει κάποιος να μπορεί να αντιδράσει όπως είπε ο συνάδελφος με εκείνα τα γραφήματα και είπαμε ότι οι περισσότερες πολιτικές χαράχτηκαν εκ των υστέρων μετά από μια επίθεση. Μετά βγήκε η πλατφόρμα και μετά επινοήθηκε και χαράχτηκε μια στρατηγική άρα χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και είπαμε στην αρχή τι γίνεται με τους μοναχικούς τι γίνεται με την επισήμανσή τους να ξέρει κανείς τι γίνεται όσον αφορά τις ε, απειλές. Έτσι να τροφοδοτείται η πολιτική για το έργο σας. Να ξέρει κανείς ποιες είναι οι απειλές. Για να γίνει αυτό χρειάζεται αυτή η θεωρία των αλλαγών που δημιουργεί αυτόν τον κύκλο πολιτικής που να είναι ενάρετος και λογικός και όχι αντίστροφο Έχουμε αυτές τις μελέτες που με χαρακτήρα πρόγνωσης και υπάρχουν εδώ κάποια κενά που θα πρέπει να αρθούν. Μετά γίνεται η χάραξη της πολιτικής, η υλοποίησή της και κατόπιν η αξιολόγηση. Να ξέρουμε αν επέδωσαν οι πολιτικές και έχουμε κάποιους στόχους που θα πρέπει να ε, επισημανθούν Επόμενη διαφάνεια. Α, αυτό μπορεί να σοκάρει για να το θέσουμε ομά. Και εδώ κάπου διαφωνούμε με τους προλαλήτες Αν κανείς θεωρήσει ότι το σημαντικό εδώ είναι η αποτελεσματικότητα, θα πρέπει η υποπτία η αξιολόγηση να γίνει όπως και στις άλλες πολιτικές. Βλέπετε εδώ όμως ότι αυτό είναι μια, ένα πολύ μικρό κομμάτι από την όλη υπόθεση. Πώς κανείς να ξέρει αν αποδίδει μια πολιτική, αν δεν τη δοκιμάσει. Να, τι λέμε στα συμπέρασματα. Αν δεν γίνει τέτοια αξιολόγηση, αν δεν γίνουν τέτοιες μελέτες πρόγνωσης, πώς κανείς ορθά τα αξιοποιήσει σε πολιτικές για να πετύχει τους στόχους που έχει καθορίσει. Τώρα, οι τελευταίες μας σκέψεις είναι, όπως είπαμε, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική υποστήριξη για τέτοιου είδου αξιολόγηση επί τη βάση στοιχείων για πολιτικές και για μέτρα. Σημαντικό, αλλά δεν ισχύει. Και έτσι να ξέρουμε τι κατεύθυνση θα πάρουμε. Άλλο. Έτσι, μια σειρά διαφορετικών σκέψεων ότι οι ομάδες των τζιχαντιστών όπως έχουμε δει και φύγει αυτό και για την ακροδεξιά είναι πάρα πολύ ευέλικτος όσον αφορά τη στρατηγική επικοινωνία. Πολλές φορές όμως δεν πάνε και καλά τα πράγματα. από πλευρά κυβερνήσεων. Δεν μπορούν οι κυβερνήσει, δεν μπορεί το κράτο να του ε, ανταγωνιστεί σε αυτό το μέτωπο. Αλλά κανεί θα πρέπει να ξέρει. Πολλά μπορούν να πάνε στραβά και είναι αντιπαραγωγικό εάν δεν έχει κανείς ως στόχο του να ανασχέσει το αφήγημα των τζιχαντιστών. Άρα θα πρέπει κανεί να έχει ένα μήνυμα ξεκάθαρο, κρυστάλλινο για το ποιος είναι, τι πρεσβεύει, τι εκπροσωπεί. Και είπαμε ότι έχουμε ως στόχο την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά κάποια στιγμή υπάρχει κάποιο είδου κόπος για πλευρά πρόληψης. Όμως, το κλειδί εδώ είναι η πρόληψη. Αυτό χρειάζεται και εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε. Μαζί με την αξιολόγηση. Να αξιολογήσουμε το πόσο αποδοτικά είναι τα προγράμματα της πρόληψης. Όμως τα αποτελέσματα δεν είναι το να ζυγιστούν ακριβώς όπως και τα μέτρα καταστολής γιατί σε αυτό το οποίο εξετάζουμε τα αποτελέσματα είναι πιο μακροπρόθεσμα και μακρόπνα. Και κατακλείδη να σας πω ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες όσον αφορά το τι γίνεται με τους πρόσφυγες και τι γίνεται με τους ετούντες που απεριφθεί η αίτησή τους και την ριζοσπαστικοποίηση. Και αυτοί μεταξύ τους τελικά αλληλοσυνδέονται, αλλοϊποστηρίζονται. Σας ευχαριστώ και τους δύο που σεβαστήκατε το χρόνο σας και μας παρουσιάσατε πολύ σύντομα τα βασικά στοιχεία και τις βασικές επικρίσεις ε, που περιλαμβάνει η μελέτη σας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντανζό και προτείνω να απαντάτε στον καθένα βουλευτή αμέσως για να είναι πιο ζωντανή η συζήτηση. Μας μένουν 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες ε, της μελέτης που περιέχει πολύ, ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και εύστοχα. Δύο πράγματα με ενοχλούν. Μεθοδολογικά, να μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας για την Ευρώπη χωρίς να έχουμε βρει Βρετανό, Γάλλο, Ισπανό, με ενοχλεί. Λέτε ότι δεν έχουμε βρει εμπειρογνώμους, δεν έχουμε θετικές απαντήσεις ακόμη τα λοιπά, αλλά πολλά θα μπορούσαν να υποθούν από τους εμπειρογνώμονες και όχι θεσμικούς απλά και μόνο από τις χώρες αυτές, αλλά σίγουρα θα είχαν συνεισφέρει ε, σημαντικά στην μελέτη. Και ένα άλλο θέμα που με ενοχλεί και το θέσατε κι εσείς είναι η μοναδοχική λύκη. Δεν μ' αρέσει η έκφραση. Χρησιμοποιεί το, το κατακόρον και πριν ε, τις επιθέσεις του 12 στην Ευρώπη. Στη Γαλλία ε, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για την υπόθεση του Μερά στην Τουλούζη το 12 και πραγματικά είναι κάτι που διαψεύδεται από όλους τους επιρρογνώμονες, ε, δικαστικούς, ε, τις υπηρεσίες, πλοφή κτλ. Γιατί μπορεί να γίνεται η πράξη από έναν δράστη, αλλά υπάρχει ο σχεδιασμός, που σημαίνει ότι παρεμβάλλονται και άλλοι. Αυτοί που ριζοσβαστικοποιούν και αυτοί που προμηθεύουν τα όπλα. Στην δίκη μερά λοιπόν τώρα. Ε, και διαβάζοντας ε, και όλη την ε, νομολογία δεν το ξέρω ποτέ να υπάρξει ένας και μόνος που να τα κάνει όλα μόνος του. Υπάρχουν ενέργειες που γίνονται και είναι εμπνεόμενες από την τρομοκρατία, από άλλους και χρησιμοποιούν ε, με ένα κουζινομάχαιρο, χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, ε, αυτοσχεδιάζουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχει ένα modus operandi διαφορετικό. Και το λέτε, υπάρχουν modus operandi με ανθρώπους που δρούν τελικά μόνοι τους ε, με αυτοσχεδιασμό και είναι και κάποιοι που δρούν με πιο επιτεδευμένο τρόπο. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε ε, ότι έχουμε να καλύψουμε ένα φάσμα 360 μοιρών, όλο το φάσμα πιθανών ε, δράσεων, τρομοκρατικών δράσεων και τρομοκρατών. Ο Αντμανί το Σεπτέμβριο το 2014 αυτό το μήνυμα λέει. Όχι το 2015 που λέτε εσείς, ήταν το Σεπτέμβριο του 2014 που λέει μανί σκοτώστε, σκοτώστε, σκοτώστε με ό,τι βρείτε μπροστά σας». Δηλαδή πάρτε ένα σφυρί, πάρτε ένα κουζινομάχαιρο και επιτεθείτε. Επίσης, στη μελέτη σα. λέτε ότι η ποινικοποίηση ανάντι των προπαρασκευαστικών ενεργειών ιδίως στο πλαίσιο της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θεωρείται αποτελεσματική από, πολλούς, από τους συμπεριλαμβανόμενους που συμβουλευθήκατε. Μα η γαλλική εμπειρία το αντίθετο ακριβώς αποδεικνύει. Από τότε που μπήκε στο γαλλικό ποινικό κώδικα η σχέση του δράστη με μια ε, τρομοκρατική ομάδα ε, ίσα ίσα. Δεν ξέρω οι δικοί σας οι και ποιοι είναι αυτοί που λένε, αλλά στην πράξη, και σας μιλώ για ένα από τα κράτη που έχει ε, τεθεί αντιμέτωπο με αυτή την ε, απειλή είναι ακριβώς ότι η ποινικοποίηση και η πρόληψη με το άρθρο του ποινικού κώδικα είναι πάρα πολύ θετική, αποτελεσματική. Το ζητάνε όλοι. Δεν είναι ένα μέτρο ασφαλείας. Ε, το ζητάνε οι δικαστικοί και το λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πραγματικά με εκπλήσουν κάποια κομμάτια της και αντί να πείτε για collection of uh, more data, λέτε improvement of uh, data. Μα και τα δύο μπορούν να γίνουν. Οι υπηρεσίε uh, πληροφοριών, η αστυνομία, η δικαιοσύνη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα. Και πρέπει να έχουν υπόψη ότι είπε και ο Επίτροπο Κίνγκ την προηγούμενη πάρα πολύ σωστό. Δεν υπάρχουν δεδομένα έτσι απόλυτα. Υπάρχουν πληροφορίες ε, από ευαίσθητες πηγές και με πολύ έτσι ειδικέ ε, διαδικασίες. Υπάρχει δικαστική συνεργασία και υπάρχουν και τα δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που είναι μια μεγάλη μάζα και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ προσεκτικά, ε, σύμφωνα με τον νόμο. Άρα ε, η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι η πανάκια, αλλά και η συλλογή ε, είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, θα ανταλλάσσουμε, αλλά πρώτα πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα. Και νομίζω ότι πιο πολύ το πρόβλημα έγκυται εκεί, στη συλλογή και όχι στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά πρέπει να απαντήσετε αρκετά σύντομα αν μπορείτε. Παρότι πολλά ήταν τα ερωτηματικά και έντονα. Παρακαλώ. Δύο λεπτά σας δίνω το πολύ. Μα αδύνατον δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος Αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Γιατί δεν μιλήσαμε με κάποιους από τους Γάλλους, Βρετανούς, Ισπανούς εμπρεγνώμονες. Δεν ήταν ότι δεν θέλαμε, αλλά Προφανώς μετά από όλες τις προσπάθειες ε, που καταβάλουμε να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους και εμείς ε, απευθείας αλλά και άλλοι συνάδελφοί μας βοήθησαν από τις χώρες μέλη και να έχουμε συνεντεύξει μαζί τους, απάρεν προφανώς και το λέω και το ξαναλέω το apparently και το προφανώς επειδή το θέμα είναι λεπτό και δεν ε, προσφέρεται για μια τέτοια ανοιχτή μελέτη, πολλοί χρησιμοποίησαν αυτό ως ε, δικαιολογία. Ότι οι υπηρεσίε τους ε, είναι απασχολημένες, έχουν πάρα πολύ φόρτο εργασίας και δεν μπορούσαν να συνομιλήσουν μαζί μα. Δεν ήμασταν εμείς που δεν θέλαμε λοιπόν. Εμείς μακάρι να είχαμε μιλήσει με όλου αυτού του συναδέλφου και με ακόμη περισσότερου. Δυστυχώ όμω αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερος δύσκολο. Και σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων, ναι, αυτό που είπα εγώ είναι ότι φυσικά υπάρχει διαφορά μεταξύ συλλογής ε, απλών δεδομένων ε, και συγκεκριμένων πληροφοριών, data και intelligence στα αγγλικά. Υπάρχει μια διαφορά στους δύο όρους και το ξέρω και από την προηγούμενη εμπειρία μου. Προσθέμενη αξία έρχεται όταν κανείς μπορεί να συλλέξει ε, τα κομμάτια του puzzle και να συνθέσει το puzzle. Η σχέση intelligence και data και αντιστρόφως. Εγώ δεν λέω ότι ανταλλαγή δεδομένων ε, είναι η χρυσή λύση, αλλά νομίζω ότι κανείς μπορεί να δει μια καλύτερη εικόνα, μια πληρέστερη εικόνα να συνθέσει τα κομμάτια του puzzle. Αυτό εντάξει είναι δύσκολο, το ξέρω σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σημειώνω ότι μπορεί να βελτιώσει την ε, αντίληψή μας για το τι συμβαίνει. Εγώ εν συντομένου με επιτρέπετε, κυρία Βαγκίνκελ, για την ε, ορολογία. Εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να προκαλεί σύγχυση η ορολογία αυτή, μοναχικός λύκος λοιπά Μπορεί να τους λένε έτσι πολύ στον τύπο, ε, στα μίντια, ε, να εκτέλεσαν την ε, πράξη μόνοι τους, αλλά σίγουρα είχαν επαφές με πολλούς άλλους. Και στο γράφημα που σας έδειξα, όταν δεν είναι δικτυωμένοι οι δράστες, ε, είναι πιο δύσκολο. Εγώ γι' αυτό σας το έδειξα το γράφημα, για να σας πω ότι οι υπηρεσίε ασφαλείας αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες γιατί βλέπουμε διαφοροποίηση των επιχειρησιακών δράσεων, και το επίπεδο της οργάνωσης των δραστών είναι διαφορετικό. Η διαφοροποίηση επίσης είναι ένα σημείο. Όλα αυτά όμως μπορούν να μας δώσουν ε, κάποια ιδέα για το τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον, σε ό,τι αφορά την ε, ποινικοποίηση των προπασκευαστικών ενεργειών. Στις συνεντεύξεις μας θέσαμε στους μενού το ερώτημα κατά πόσον χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία για να μπορούν να προχωρούν σε έρευνα ή δίωξη. Και μας είπαν όχι, δεν θέλουμε, υπάρχει αρκετή νομοθεσία και είναι αποτελεσματική. Και κάποιοι είπαν ότι ούτε καν χρησιμοποιούν όλα τα νομοθετήματα που είναι διαθέσιμα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Άννα Γκόμες, για ένα λεπτό όμως. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Ένα λεπτό. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι σημαντικό να έχουμε να παρουσιάσουμε κάποιες επιτυχίες για την αποτροπή και καταπολέμηση της ρίσος παστικοποίησης. Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση με τι νοφιλελεύθερε πολιτικές και τη γλώσσα και το αφήγημα των κυβερνήσεών μας, διότι είναι τεράστια κοινωνική επένδυση που απαιτείται. Και αυτό δεν έγινε βέβαια. Και ούτε και θέλουν να το κάνουν. Δεύτερο ερώτημα. Η σχέση των δημοκρατικών ομάδων με το συνοριακό έγκλημα, διακρατικό έγκλημα. Συμφωνώ. Δεν βλέπετε επίση ότι με αυτή τη διασύνδεση Δεν είναι μόνο τα όπλα και το φρολικό έγκλημα και τα ναρκωτικά, αλλά όλο το σύστημα. Το σύστημα χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα χρήματος. Για τις εγκληματικές ομάδες και τις τρομοκρατικές ομάδες. Στα κράτη και στο χρηματοοικονομικό, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με τα think tank, τα bitcoin και όλα αυτά που δεν καλύπτονται καν, όπως είπατε κι εσείς από την οδηγία αυτή. Μήπως εκεί δεν θα έπρεπε να ξυπνήσουν οι κυβερνήσεις για να ελέγξουν και να συγκρατήσουν αυτό το σύστημα που είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Απάντηση, ακούστε, το πολιτικό κλίμα φυσικά και επηρεάζει σημαντικά τις, τους πόρους και το πώς δαπανώνται αυτοί. Και κατά πόσο υπάρχει επιθυμία να επενδύσει κανείς σε ιστορίες επιτυχίας ή αν το κλίμα ε, είναι κάπως ε, κλίμα τρομοκρατίας. Εγώ δεν είμαι υπέρ βέβαια του δεύτερου και ελπίζω να έχω υπόψη μας μια συνολική προσέγγιση και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Το επόμενο ερώτημα για τη σχέση, τη διασύνδεση των δύο. Πράγματι, με τη διασταύρωση και διασύνδεση αυτών των τομέων μπορούμε να αναλύσουμε και να δούμε τι εξελίξει έχουν παραδείγματο χάρη στο δεσυνοριακό διεθνέ έγκλημα. Μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό για τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Αντί να το δούμε και των υστέρων, να προκαταλάβουμε τι εξελίξει. Ότι μπορεί το οργανωμένο έγκλημα να είναι πολύ ελκυστικό ε, και μπορεί να αξιοποιηθεί από του τρομοκράτε. Και έτσι μπορούμε να προλάβουμε ενδεχομένω Μάιτε Παγάθα Ουρτουντούα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Γιατί είμαστε εδώ, γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ασφάλειας και έχουμε την έννοια της Ένωσης ε, Ασφαλείας κατά κάποιο τρόπο. Και θα πρέπει να υπάρξει προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην ε, μελέτη που μας παρουσιάσατε είναι μια της μελέτης, στη σελίδα 32 κάτι για τα στατιστικά που λέτε, μιλάτε για τον αριθμό των θανάτων από το 2001 έως το 2015, θα θυμάτων τρομοκρατίας. Και αυτό που βλέπω εγώ, ότι δεν υπάρχει, και χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ. Για Ευρωπαίους δεν έχουμε στοιχεία για την περίοδο αυτή που έχασαν τη ζωή του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Γιατί σα το λέω αυτό, γιατί λέτε ότι πρέπει οι μελέτε μα να είναι στραμμένες προς το μέλλον. Ναι, αλλά πρέπει να αντιπαραβάλλετε τα στοιχεία και τα στοιχεία αυτά να είναι ποιοτικά. Γιατί μου δίνετε την εντύπωση ότι δεν έχουμε ακόμα μία βάση δεδομένων ευρωπαϊκή. Και υπάρχει και ένα θέμα. Ενιολογικό θέμα σχεδιασμού. Ποιο θεωρείται θύμα τρομοκρατία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ειρηνευτικές αποστολέ, ε, άμαχος πληθυσμό ε, ή άλλοι. Όλα αυτά δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Επίση, αν δεν έχουμε καλά στατιστικά στοιχεία για τα θύματα τη τρομοκρατία, δεν μπορούμε να ε, έχουμε και τη σωστή αντιμετώπιση. Τι γίνεται με τι νομοθεσίε, αν ούτε αυτό το έχουμε μελετήσει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι ένα δύναμο σημείο της έκθεσης ο διευθυντής των, του Κέντρου Μελετών, Αμυντικών Μελετών, ο Ισπανός ε, στρατηγός Βερεστέρος λέει ότι ε, σημαντικό στοιχείο στην καταπολέμηση και για ενίσχυση της ε, των κοινωνιών είναι ε, το να δούμε τι γίνεται με τα θύματα. Γι' αυτό λέω, θα έχετε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για να μην υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Το 2001, 120 Ευρωπαίοι είχαν χάσει τη ζωή της την 11 ε, Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αυτά τα χρόνια που εσείς λέτε υπάρχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω, θύματα Ευρωπαίοι σε επιθέσεις τρομοκρατικές και δεν τα αναφέρετε. Επίσης ε, μου κάνει τρομερή εντύπωση που οι Ισπανικέ αρχέ ασφάλεια δεν σα έδωσαν τι πληροφορίε. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Πρόεδρο, ένα λεπτό. Δίνω... Ε, έπρεπε να τελειώσουμε στι 5.30, αλλά θα δώσω 5 λεπτά παραπάνω για την άλλη δύο συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Λοιπόν, μία απάντηση από εσά ένα λεπτό. Και έχω και τους ε, ομιλητές που έχουν γραφτεί Λοιπόν, ένα λεπτό εσείς, οι συνάδελφοι, και μετά κλείνουμε. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο κανείς να φτιάξει τη δική του βέση δεδομένων, οπότε και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό κατά την μελέτη. Και μετά προσπαθήσαμε, βέβαια, άκουσα τι είπατε όσον αφορά το Πανεπιστήμιο του Maryland. Ε, είναι αυτό είναι παγκοσμίω αναγνωρισμένο ότι έχουν πάρα πολύ καλή βάση και χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα με πολλούς τρόπους. Και εμεί έχουμε εδώ πέρα κάποια δεδομένα ανά αναπεριοχή, ανά τη ΣΕΛΑΚ. Μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία, Βεβαίω και μπορείτε να ενημερωθείτε και έτσι να έχετε μια πληρέστερη εικόνα του τι ισχύει. Όσον αφορά την νομοθεσία, είπατε ότι χρειαζόμαστε ένα ίδρυμα ευρωπαϊκό να συλλέγει αυτά, να κάνει ανάλυση. Ε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Έχουμε τώρα την Europol και άλλες υπηρεσίες. Ναι, δεν έχουμε τώρα απόφαση, δεν έχουμε δεδομένες ε, εκθέσεις και μελέτες σε τακτέ διαστήματα. Γίνονται προσπάθειες από πολλά κρατή-μέλη και μας ζήτησε η Λίμπη να διαλέξουμε ποιες χώρες για να κάνουμε μελέτη. Διαλέξαμε 7 και έτσι γίνεται η εφαρμογή αυτής της απόφασης. Pardon. Yann Philippe pour une minute. Äh, Φιλίπ. That for the future all the coordinators will have the same opportunities. Όλοι οι συντονιστές θα πρέπει να είμαστε ε, ίσοι. Δεν ισχύει αυτό. Να το κάνουμε αυτό στο μέλλον. Όλοι οι συντονιστές ίδιο χρόνο για να υποβάλουμε τις ε, ερωτήσεις στους προσκεκλημένους. Τέλος πάντων, επί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μελέτη και νομίζω θα πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία αναδύθηκαν ιδίω ότι θα πρέπει να δούμε για καλύτερη εφαρμογή των προβλεπωμένων μέτρων. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα το βλέπει σοβαρά το θέμα. Να βελτιωθούν τα υπάρχοντα νομοθετήματα. Παρά όσον αφορά τα δεδομένα, ε, βέβαια και καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να επεκταθούν τα μέτρα για περισσότερη συλλογή δεδομένων ή συλλογή περισσότερων δεδομένων απλώς. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Χρειάζεται όμως βελτίωση για την ανταλλαγή των δεδομένων. Εκεί να προσπαθήσουμε, σε αυτό το μέτωπο και όχι στο θέμα της συλλογής αυτών. Είναι όλοι αυτοί οι μοναχοί λύκοι, πάντοτε υπάρχουν διασυνδέσεις. Και άρα θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά οι αρχές και να αξιοποιούν τις παρασχεθήσεις πληροφορίες. Κύριε Φανόρντεν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να δείξω αυτό το λεπτό θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Και δεν μιλώ για αυτούς που είναι τρομοκράτες, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε μεγάλης κλίμακας μετανάστευση, μεγάλης κλίμακας ε, κύμα ετούν των άσυλο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι επομένω όλο ένα και πιο δύσκολο αυτοί να ενταχθούν κοινωνικά. Όλο ένα και περισσότερο εξαντλούμε τις δυνατότητες των διοκτικών αρχών. Είναι όλο ένα και περισσότερο αυτοί που πρέπει να παρακολουθούνται. Δεν προκάνει η αστυνομία. Ε, άρα, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για πέστε με την άποψή σας. Et enfin, Eva Jolie, pour conclure. Eva Jolie, τελευταία, για να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι στη μελέτη αυτή Ελείπει μια πηγή εύκολης πρόσβασης, η δικαστική. Στο Παρίσι έχουμε ένα δικαστήριο ειδικό για θέματα τρομοκρατίας και για αυτούς που τους χρηματοδοτούν. Η δικαστή υπεύθυνη είναι η Ζαμπέλ Πρεβόντε Πρέ. Συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι προσβάσιμες. Ξέρουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μιλάμε για μοναχικούς λύκους. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι χρηματοδοτούν την προετοιμασία μιας τρομοκρατικής πράξης και οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού παρουσιάζουν με πάρα πολύ μεγάλη ενάργεια την προετοιμασία μιας τέτοιας τρομοκρατικής ενέργειας. Και νομίζω ότι ε, θα μπορούσαμε αν τη συναντήσουμε, αν τη συναντήσετε, να σας δώσει την ουσία των σκέψεών της και να σας μεταφέρει και την ουσία των αποφάσεών της, σαν παράδειγμα. Ένας ε, οι μητέρες ε, δεν επηρεάζονται σαν παράδειγμα μόνο για την ευημερία του παιδιού τους όταν το χρηματοδοτούν, αλλά ταυτόχρονα και για τη δική τους θέση στον παράδεισο, γιατί τα παιδιά λένε στις μητέρες ότι αν σκοτώσουν ένα άπιστο θα έχουν και οι μητέρες των τρομοκρατών μια θέση στον παράδεισο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, λέει η κυρία Γκρισμπέκ. Επικοδομητική η πρόταση και καλό θα ήταν να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση. Σας δίνω το λόγο πάρα πολύ σύντομα να δώσετε μια πολύ σύντομη απάντηση και να κλείσει η συζήτηση εδώ. Θα είμαι σύντομος για, τα, για τις τράπεζες δεδομένων Είδαμε ότι πολλοί που εμπλέκονται στη δίωξη της τρομοκρατίας δεν θέλουν να διευρυθούν οι δυνατότητες για συλλογή στοιχείων και δεδομένων. Αλλά ταυτόχρονα είπαν ότι υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά των δεδομένων που είναι πολύ ωφέλιμα. Σαν παράδειγμα, συλλογή στοιχείων από πλευράς των στρατιωτικών αρχών για πληροφορίες από τα πεδία μάχης διαμετρήματα όπλων κτλ. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία σίγουρα μπορεί να βοηθήσουν ιδιαίτερα στον εντοπισμό αυτών οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επανέλθουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Και να δούμε τη σχέση που έχει αυτό το θέμα με την μετανάστευση, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Πάντως, η βασική ιδέα δεν είναι να συλλέγουμε περιτότερα συστήματα δεδομένων, αλλά να χρησιμοποιούμε τα ήδη υπάρχοντα. Για τα θέματα της μετανάστευσης πάλι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς που παρουσιάζουν πράγματι ενδιαφέρον. Ε, να υπάρξει κατάχρηση των μεταναστευτικών ραών από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, σαν παράδειγμα. Από την άλλη είναι σαφές ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα αναμονής για τη χορήγηση ασύλου πολλές φορές περνούν μήνες για να μην πω χρόνια χωρίς καμία θα έλεγα ελπίδα για το μέλλον και προοπτική για το μέλλον κάτι το οποίο τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στους στρατολόγους των τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε να ενισχύσουμε τις ομάδες αυτές, να τις καταστήσουμε πιο ανθεκτικές στις πιέσεις των στρατολόγων τους. Ελπίζω ότι η δική σας επιτροπή το συγκεκριμένο θέμα θα το λάβει σοβαρά υπόψη. Υπάρχει και το θέμα επίσης ε, συνεντεύξεων και επαφών με ανθρώπους που είναι πηγές πληροφοριών. Γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά να πούν και δεν είναι σε θέση να τα πούν σε σωστό χρόνο και με σωστή μορφή, κάτι το οποίο δημιουργεί δυστημία και σε αυτούς που επεξεργάζονται τα στοιχεία εκ των υστέρων. Ελπίζω λοιπόν τα στοιχεία αυτά να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει και να τα εκμεταλλευτεί έγκαιρα. Θέλω πάντως να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας περαιτέρω για άλλες ερωτήσεις. Τελειώσαμε εμείς τη δουλειά μας για την έκθεση αυτή, αλλά για το Ινστιτούτο μας τα θέματα αυτά είναι πάντα στην επικαιρότητα και είμαστε στη διάθεσή σας ε, να συνεισφέρουμε σε ερωτήσεις σας ή να κάνουμε άλλες έρευνες αν τις χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ λέει η κυρία Γκρισμπεκ, τους δύο ομιλητές μας που έκαναν μια παρουσίαση την οποία θελήσαμε να είναι αρκετά συμπυκνωμένη και ταυτόχρονα υπέστησαν το παιχνίδι των ερωταπαντήσεων. Πολλές φορές οι ερωτήσεις ήταν αμεσότατες, αλλά δώσατε απαντήσεις ζητώντας και από τους συναδέλφους να συνεχίσουν το διάλογο μαζί σας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν για τα μέλη γιατί ξεπεράσαμε την κανονική διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής μας. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να σέβεστε στο μέλλον το χρόνο ομιλία σας για να υπάρξει μια πλήρης ισοτιμία ανάμεσα στους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ όλους μια πρακτική ενημέρωση σχετικά με την επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας 26 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο από τις 9 μέχρι τις 12. Θα πάρετε την ημερήσια διάταξη εγκαίρως μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ παρακαλώ όμως τους συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα έτσι ώστε να ξεκινήσει η δική μας συνεδρίαση Άμεσα σχεδόν. Λοιπόν, όσοι πρέπει να φύγουν, παρακαλώ να το κάνουν πολύ γρήγορα και να παραμείνουν αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν.